Right. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν όλους. Ε, νομίζω ότι έχουμε αρκετά μέλη στην αίθουσα ε, για να μπορούμε να ξεκινήσουμε για τα σημαντικά κυρίως θέματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω το εξής. Ε, έχουμε μπροστά μας την έγκριση της ημερήσιας διάταξης και Νομίζω ότι έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μα. Ε, αφαιρέθηκε ένα θέμα από τη μέση διάταξη, ο κύριο Τρισέ, γιατί ήταν εδώ τη Δευτέρα. Και έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με την Ευρωπαϊκή ε, Ρυθμιστική Αρχή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου. Έτσι λοιπόν ε, φαντάζομαι θα μπορούμε να τη βρίσκουμε το χρονοδιάγραμμα και ελπίζω αυτοί που έχουν προγραμματίσει να έρθουν για συγκεκριμένα θέματα να έρθουν στην ώρα τους. Από ό,τι βλέπω κανείς δεν διαφωνεί στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Τώρα, ανακοινώσεις της ε, Προέδρου. Έχουμε πρώτα απ' όλα το εξής. Να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής μας θα λάβει χώρα στις 12 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Στρασβούργο, στις 7 η ώρα το βράδυ και ε, θα σας σταλεί έγκαιρα η ημερήσια διάταξη. Ε, το δεύτερο που θέλω να πω είναι να σας ε, ενημερώσω λιγάκι για την ε, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της EBRD που έγινε χτες το βράδυ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Ε, είχαμε την πρώτη ανάγνωση στο Συμβούλιο το οποίο είχε κάποιες επιφυλάξεις για το κείμενο το οποίο είχαμε διαπραγματευτεί σχετικά με τον ορισμό των φορολογικών παραδείσων. Ελπίζω λοιπόν ότι τελικά το αποτέλεσμα θα μας ικανοποιήσει. Θελήσαμε να συμπεριλάβουμε έναν ευρύτερο ορισμό από αυτόν που αναφέρει ο ΩΣΑ. Γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε το αποτέλεσμα και ελπίζουμε να ε, ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ε, ψηφίσουμε στην, στις 2 Σεπτεμβρίου. Και ε, θα σας ενημερώσω σχετικά με τις ε, αντιδράσεις της ε, Προεδρίας σχετικά με, το, με τα θέμα ή τα θέματα που εκκρεμούν. Αυτά είχα να σας πω ως ανακοινώσεις Προέδρου και τώρα λοιπόν πάμε στον, ε, στο σχέδιο προεπολογισμού του 2012 στην εξέταση των τροπολογιών από τον εισηγητή που είναι ο κύριος Λούτβιξον ε, δεν αναφέρεται μπροστά στα χαρτιά μου, αλλά ξέρω ότι είναι ο κύριος Λουτρίξον γιατί έχει λάβει το χώρο επανειλημμένα κατά το παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Γνωρίζετε ότι θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα επί του προϋπολογισμού. Υπάρχουν λοιπόν τέσσερα σημεία ε, που τα βρίσκουμε σημαντικά. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό η νέα εποπτική αρχή να έχει αρκετού πόρου για να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Η φιλοδοξία του Συμβουλίου να περιορίσει τις, ε, τα ποσά που αναφέρει η Επιτροπή, αυτή δεν είναι και πάρα πολύ καλή ιδέα. Εμείς λοιπόν θα θέλαμε οι ε, εποπτικές αρχές να λειτουργήσουν με βάση τους ε, προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για μας ε, είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε επί της αρχής, δηλαδή οι υποπτικές αυτές αρχές να έχουν ε, να και με περαιτέρω πόρους. Και δεύτερον, χρειαζόμαστε ένα είδος διοικητικού μηχανισμού για να στηρίξουμε το σύστημα και για να συνεχίσουμε το δρόμο που έχουμε ήδη χαράξει Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις, να αυξήσουμε τη διαφάνεια και τον έλεγχο, ε, να είμαστε σίγουροι ότι εφαρμόζονται οι κανονισμοί ε, και αυτό ελπίζουμε να συμβάλλει στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Κατόπιν πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για να πάψει πλέον, να πάψουν να υπάρχουν αυτή η φορολογική παράδοση. Ε, νομίζω ότι αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας και είναι σημαντικό για μας ε, να συνεργαστούμε στο πλαίσιο του προγράμματος ε, Φισκάλης, ε, να υπάρχει διεθνή συνεργασία επί του θέματος. Κατόπιν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα πρόγραμμα που λειτουργεί πάρα πολύ καλά, το CEP, το οποίο επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν καλύτερη πρόσβαση στο κεφάλαιο. Ε, το, ε, κεφάλαιο, το Συμβούλιο βέβαια επιθυμεί να προβεί σε εξοικονομήσεις, αλλά ε, το να έχουμε πολύ χαμηλό επίπεδο πιστώσεων αυτό δεν είναι σωστό. Το πρόγραμμα προσφέρει εργαλεία ε, τα οποία χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε ε, το δυναμισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, εξακολουθούν να μην έχουν ε, ανακάμψει μετά την οικονομική κρίση του 2008 και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σκιώδη Συγήτρια για την πολύ καλή συνεργασία. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. καταρχήν λοιπόν η Άστριτ, η πρώτη Σκιώδη Συγήτρια.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 Θα ήθελα να πω ότι συμφωνούμε απολύτως με τον εισηγητή. Και χθε όλοι όλοι οι εισηγητές συμφωνήσαμε για τις συμβαστικές τροπολογίες. Απλώς και μόνο θα ήθελα να πω ότι είμαστε υπερήφανοι διότι δημιουργήσαμε αυτούς ε, τους εποπτικούς οργανισμούς που είναι η κατάλληλη λύση για να μπορέσουμε να ασκήσουμε την εποπτεία και τον έλεγχο που θέλουμε. Εάν όμως αρνηθούμε τα κατάλληλα κονδύλια για να κάνουν σωστά την εργασία τους, θα ανακόψουμε την πορεία τους. Πράγμα το οποίο θα χαροποιήσει κάποιους οι οποίοι δεν ήθελαν να δημιουργηθούν αυτοί οι εποπτικοί οργανισμοί. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τις πιστώσεις, τα κονδύλια που δίδονται σε αυτούς τους οργανισμούς. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Στη μικρή μου χώρα, το Λουξεμβούργο. Ο έλεγχος των οικονομικών υπηρεσιών, η δημοσιονομική εποπτεία αν θέλετε, Απασχολεί περίπου 400 με 500 άτομα. Και στην Ευρώπη ο αντίστοιχος τραπεζικός πεπτικός οργανισμός θα απασχολήσει 60 άτομα. Ίσως θα μπορείτε να πείτε στους ε, αρχηγούς κρατών σας ότι ε, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να γίνουν οικονομίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούμε εμείς αύξηση των πιστώσεων. Όσον αφορά τις άλλες συμβαστικές τροπολογίες, συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όλε. Ευχαριστώ. Ο Καρλ Άγγλοντ είναι σκέδης αλλά δεν μπορεί σήμερα να είναι συνεδρίαση. Ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα της ε, Φινλανδίας που ίσως δεν είναι μία από τις πρωταγωνίστρες χώρες στην συζήτηση αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει εκστρατεία για το προεδρικό αξίωμα στην Φιλανδία και αυτό δεν είναι εδώ συνάλφος. Συμφωνήσαμε τις ε, τροπολογίες συμβαστικές, δεν υπάρχουν γενικότερες δυσκολίες, αλλά μπορώ και εγώ να συμφωνήσω και με την Άστριντ όσον αφορά την υποστήριξή μας προς αυτή την Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας. Εάν μειώσουμε τα κονδύλια δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Συγχρόνως όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι όταν λέμε το πιο σημαντικό θέμα συζήτηση είναι οι αριθμοί, εγώ θα έλεγα ότι η ποιότητα είναι ακόμη πιο σημαντική. Η ποιότητα του εργασίας που θα επιτελέσουν αυτά τα άτομα για τον έλεγχο. Θέλουμε ένα προπολογισμό ποιοτικό και προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα. Συμφωνούμε όλοι. Βεβαίω είναι σημαντική αρχή, αλλά νομίζω ότι είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο σημαντική, η ποιότητα. Και η περισσότερη εποπτική δουλειά θα γίνει στα 27 κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ο σωστό συντονισμό. Θα έλεγα λοιπόν ότι η ανταπόκριση συμβουλή δεν είναι πολύ ε, καλή. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε και τη Eurostat. Διότι η στατιστική είναι σημαντική και ξέρουμε ότι υπήρχαν προβλήματα στο παρελθόν. Η ποιότητα των δεδομένων της στατιστικής είναι κάτι το απαραίτητο. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια στα πλαίσια του προπολογισμού για να βελτιωθούν τα πράγματα. Η Άλντε σας ε, ε, ευχαριστεί συνάδελφε Ούλα για την εξαιρετική δουλειά που επιτελέσατε. Ευχαριστώ. Κανένα άλλο δεν ζητά το λόγο. Ο Σβέν. Πάρα πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδες εισηγητής. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων. Συμφωνούμε με τον εισηγητή και συμβαστικέ τροπολογίε, απλώ θα ήθελα να τονίσω ότι για ε, αυτού του οργανισμού οργανισμούς η πρόταση του Συμβουλίου να υπάρξουν περικοπές σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής είναι κάτι το οποίο βρίσκουμε παράδεκτο. Εάν δείτε ποια είναι το προσωπικό που προβλέπονται και σε σχέση και το τι γίνεται στους εθνικούς οργανισμούς εποπτείας, είναι παράλογο όλα αυτά θέλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε την καλά την τάλληλη νομοθεσία για να εξοικονομήσουμε χρήματα και αν θέλουμε να το πράξουμε αυτό θα πρέπει και να γίνει κάτι σε εθνικό επίπεδο τι ε, εθνικοί οργανισμοί. Στη χώρα μου υπάρχουν 1.700 άτομα που δουλεύουν στον ε, αντίστοιχο οργανισμό, τον Μπάφιν. Και στην χώρα μου κανείς δεν ξέρει αν αυτό είναι σωστό, είναι απαραίτητο. Στη Γερμανία έχουμε περισσότερα 7 ε, άτομα, 7 φορέ περισσότερα άτομα από ότι αυτό το οποίο προβλέπεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Το ίδιο συμβαίνει στον Πανευρωπαϊκό αυτό Οργανισμό εποπτεία. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλε χώρε, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν πρόκειται εδώ για κατασπατάληση χρήματος. Χρειαζόμαστε το κατάλληλο προσωπικό, τον κατάλληλο οργανισμό και τον κατάλληλο συντονισμό. Γι' αυτό θα πρέπει, σωστά όπως λέγεται, να ξεπεράσουμε την ε, πρόταση της Επιτροπής, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο ζήτησε ο ίδιος αυτός ο οργανισμός. Δεν είναι κάτι που εμείς εφήβραμε, είναι κάτι το οποίο ζήτησε ο ίδιος ο οργανισμός για να μπορέσει να λειτουργήσει και νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς να είμαστε ε, σύμφωνοι με αυτά τα οποία πρότεινε και η δική μας Επιτροπή Προπολογισμών και να ψηφίσουμε σχετικά, την σχετική πρόταση η οποία είναι πολύ λογική. Ευχαριστώ. Πόρτας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ Πρέπει να πω ότι γενικά συμφωνώ με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις οι οποίες υπευλήθηκαν και ιδιαίτερα με όσον αφορά τα θέματα που αφορούν την καταπολέμηση της απάτης φοροδιαφυγής, αυτά τα οποία ελέγχθη για την υπηρεσία στατιστικής και με την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εποπτείας. Έχω δύο ερωτηματικά. Ο Γκίλγουντ, ο συνάδελφος, είπε ότι τα νούμερα, τα οποία αριθμοί που προτείνονται για αυτές του οργανισμούς εποπτείας είναι αυτά τα οποία ζήτησαν οι ίδιοι αυτοί οι οργανισμοί. Εγώ είχα κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά το κριτήριο το οποίο ακολουθήθηκε για την πρόταση αύξησης ε, σε σχέση με την πρόταση Επιτροπής. Τώρα όμως κατάλαβα ποια είναι η ουσία του προβλήματος και κατάλαβα που προέρχονται αυτοί οι αριθμοί. Ούτως ή άλλως πρέπει να πω ότι υπάρχει μια πρόταση με την οποία δεν συμφωνώ η πρόταση με το πρόγραμμα πλαίσιο για την καινοτομία και την ε, ανταγωνιστικότητα. Η πρόταση του εισηγητή είναι να υπάρξει αύξηση μέρους 70 ε, εκατομμυρίων πιστώσεων για τις πληρωμές. Δεν γίνεται λόγος όμως για τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Έχω αμφιβολία. Διότι νομίζω ότι αυτή η τροπολογία του 2012 συζητείται σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι πραγματικά αρνητικό γενικότερα. Για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε τις πληρωμές θα πρέπει να έχουμε και τα αντίστοιχα ποσά και στις υποχρεώσεις. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, εάν δεν συνδεθούν τα διαθέματα, τι κάνουμε. Ζητούμε περισσότερες πληρωμές, αλλά δεν έχουμε εξασφαλίσει τις υποχρεώσεις. Θα πρέπει λοιπόν οι αυξήσεις να γίνουν ε, και στα δύο αυτά ε, κομμάτια για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουν και θα είναι πραγματικές. Ευχαριστώ. Αστρίντ, θες να απαντήσεις ή όχι. Θες και πάλι το λόγο. όχι, όχι, όχι. Ό,τι είχα να πω το είπα. Είπα ότι συμφωνούμε. Ας μην χάνουμε χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη. Εντάξει, όλοι. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι δεν έχω να προσθέσω τίποτε, δεδομένου ότι όλες οι συμβιβαστικές απόψεις συμφωνούν. Προσπαθήσαμε να βρούμε σημεία σύγκλησης. Ξέρουμε ότι η οικονομική κατάσταση δεν είναι εξαιρετική, υπάρχουν μεγάλες ασάφειες και ερωτηματικά και εγώ λέγω ότι πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε τις σωστές επιλογές για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ όλους όσους συνεισέφεραν στη συζήτηση και στη συμφωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σήμερα το απόγευμα θα ψηφίσουμε και προχωρούμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση στην εσωτερική αγορά. Συντάκτρια η Σοφία Οκονή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχηθώ στους συναδέλφους καλή επάνωδο. Η έκθεση αυτή για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση στην εσωτερική αγορά είναι το θέμα μου και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες για να εμπλουτιστεί αυτή η γνωμοδότηση. Ο στόχος μας με τις συμβαστικές τροπολογίες να έχουμε ένα συνεκτικό κείμενο και χάρη στις αποτελεσματικές και επικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων με τους συναδέλφους νομίζω ότι υλοποιήσαμε το στόχο μας. Πριν να ε, περάσω στις γενικές γραμμές θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια οικονομικά στοιχεία για το τομέα αυτό. Ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών σε απευθεία σύνδεση έχει έσοδα τα οποία το 2008 ξεπέρασαν τα 6 δις η Ευρώπη είναι το 45% της παγκόσμιας αγοράς και ο τομέας αυτός τυχερών παιχνιδιών σε επευθείας είναι αποτελεί το 7,5% των τυχερών παιχνιδιών γενικότερα και θα είναι τομέας που το 2013 θα διπλασιαστεί, θα είναι το 15%. Θα πρέπει λοιπόν να τον εξετάσουμε μεγάλη προσοχή. Όπως πάρα πολλοί συνάδελφοι υπογράμμισαν όταν κατέθεσαν τροπολογίες θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη χρησιμοποίηση των τυχερών παιχνιδιών απευθείας από ε, παράνομα δίκτυα και παίκτες. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων και των ε, εποπτικών αρχών και της Κομισιόν και της Europol πάρα πολύ καλή συνεργασία και μεγάλο συντονισμό. Θα πρέπει να μπορέσουμε να θεσπίσουμε κανόνες διαλειτουργικούς για να μπορούμε να δούμε πώς θα καταπολεμήσουμε την απάτη, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και οποιαδήποτε προσπάθειες παράνομων δραστηριοτήτων, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε πρώτα απ' όλα την επιτύχουμε να έχουμε καταχώρηση όλων των παράνομων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να έχουμε τα μέσα που θα μας επιτρέψουν να καταπολεμήσουμε τις ε, παράνομη προσφορά τέτοιου είδους τριχερών ε, παιχνιδιών και να αφήσουμε την ελευθερία στα κράτη-μέλη να δούνε ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ρυθμίσουν τα στοιχήματα απευθείας και τα τυχερά παιχνίδια ή απαγορεύοντάς τους ή ε, υποβάλλοντάς τα στο καθεστώς του εθνικού μονοπωλίου ή με άλλους τρόπους για να καθορίσουν νόμιμους τρόπους λειτουργίας αυτού του τομέα. Και θα πρέπει για την προστασία των καταναλωτών να έχουμε ελάχιστα στάνταρ, αλλά και για θέματα ευθύνης και νομιμότητας να νομολογήσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς έχει επίσης το θέμα της εξάρτησης από τέτοια παιχνίδια και πώς θα προστατεύσουμε από αυτά τα παιχνίδια και τους ε, ε ανήλικους. Ο Θεόδωρος Κυλακάκης πρότεινε να γίνουν μελέτες ε, για το θέμα αυτό στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική η πρότασή του και θα πρέπει να προβλέψουμε και δυνατότητες αυτοελέγχου. Κατά την ε, εγγραφή ε, απευθείας με, τρόπο, με, στον, με ηλεκτρονικό τρόπο αυτών οι οποίοι θέλουν να παίξουν τέτοιους παιχνίδια. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά στοιχήματα και θα πρέπει να μπορέσουμε να ευνοήσουμε και την ανταλλαγή απόψεων τη σωστή μεταξύ αυτών που κάνουν τα στοιχήματα των δημοσίων αρχών και των αθλητικών ε, υπευθύνων. Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι η κινητήριο δύναμη για τη διευθέτηση του προβλήματο αυτό. Διότι αν υπάρχουν εθνικά διακυβεύματα, η συνεργασία θα πρέπει να είναι διακρατική. Θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε και μία κοινή ε, κοινό ορισμό των ε, αδικημάτων, παραπτωμάτων και απατών και θα πρέπει με την βοήθεια των φορέων για τα στοιχήματα και των αθλητικών αρχών να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταπολεμήσει την απάτη στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει λοιπόν να διαδραματίσει ρόλο συντονιστικό στον οποίο το νέο άρθρο 165 της συνθήκης αναφέρεται και θα ήθελα να πω ότι τα στοιχήματα, και είναι σημαντικό αυτό κύριε Πρόεδρε, να λάβουμε υπόψη ότι τα τυχερά παιχνίδια και τα στοιχήματα δημιουργούν κέρδη τα οποία αναδιανέμονται στον ε, χώρα και είναι μια πηγή χρηματοδότησης. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιό να μελετήσει τα μέσα που θα επιτρέψουν αυτό το χρηματοδοτικό μέσο να το διευθεντήσει από νομικής απόψεως ώστε να υπάρχει ακαιρεότητα και στην ε, τομέα του επαγγελματικού αλλά και του ε, αθλητισμού εκτός επαγγελματικών τομέων. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την συντάκτρια για τη συνεργασία της. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Είναι πολύ καλό να γνωρίζουμε ότι όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν τις ίδιες πεπιθήσεις στο θέμα των στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών και το γεγονός ότι υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι αλλά και πολλές ευκαιρίες στα στοιχήματα. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν φέρει τροπολογίες που έχουν να κάνουν με θέματα προστασίας των καταναλωτών και πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλες οι τροπολογίες μας έχουν ληφθεί υπόψη στους συμβιβασμούς και ως αποτέλεσμα ε, ε πάρα πολύ με τον τρόπο χειρισμού των προτάσεών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Κυρία Κόνη, έχει ξεκινήσει μια πολύ επικοδομητική συνεργασία με τους σκιώδεις στις τοπολογίες και πιστεύω ότι έχουμε ε, μια ενδιαφέρουσα σειρά τροπολογιών και ε, ε των οποίων πρέπει να ψηφίσουμε. Ε, Ζητήμα από την Κομισιόν να διερευνήσει εάν το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι αναγκαίο στην Ευρώπη και θα είναι ενδιαφέρον να το εξετάσουμε αυτό. Τούτου λεχθέντος, επιγραμμικά online σημαίνει ότι εξορισμού είναι διακρατικά, διασυνοριακά και θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία. Η επικουρικότητα ε, φυσικά είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρξε απόφαση από το δικαστήριο που αναφέρει ότι είναι μια υπηρεσία τα τυχερά παιχνίδια, τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με κάποιους κανόνες της παροχής υπηρεσιών. Θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες. Ε, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος ως αποτέλεσμα των ε, κανόνων που έχουν ε, συμφωνηθεί από την Ένωση έχει και περιορισμούς στον τομέα των στοιχημάτων σε απευθεία σύνδεση. Και είναι σημαντικό ότι αυτή ε, οι περιορισμοί θα είναι ε, λόγοι να θέσουμε πιέσεις. Ε, θα πρέπει να δικαιολογήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την συμπεριφορά της και να εξηγήσει γιατί έχουν ληφθεί αυτά τα μέτρα και θα πρέπει να δικαιολογήσει ότι είναι αναλογικά ως προς τους στόχους. Δεν είμαστε υπέρ μιας απαγόρευσης, γενικής απαγόρευσης των απευθείας τυχερών παιχνιδιών είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθηθούν και είναι πολύ δύσκολο να επιβληθεί με τέτοια απαγόρευση. Πρέπει να ε, δούμε ότι συμμορφώνονται με τις επιθυμίες ε, ε, αυτών που θέλουν κανονικά να συμμετέχουν σε αυτά τα παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση. Ε, θα πρέπει βέβαια να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα χρήματος. Συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια σε αυτό το θέμα και ε, υποστηρίζουμε επίσης την δομική συνεργασία ανάμεσα στους εθνικούς ρυθμιστές. Είναι ένα θέμα το όπου θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες ανταλλαγές όπου θα μπορούν οι χώρες να δουν ποια είναι τα προβλήματα σε κάθε χώρα και να δουν πώς μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Ε, και μπορούμε να μάθουμε πολλά σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε ακούσει για την προστασία των καταναλωτών, είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό, θα πρέπει να τα κρατήσουμε αυτά τα στοιχεία. Τώρα, αν ε, μιλάμε ε, τώρα και για τον αθλητισμό θα πρέπει να το εξετάσουμε, αλλά όπως έχει ελεγχθεί είναι κάτι παραπάνω από αθλητισμός. Ένα μεγάλο μέρος των λεφτών που είναι ως έσοδα χρησιμοποιούνται για καλούς σκοπούς. Δεν θέλουμε αυτή την πηγή χρηματοδότησης να σταματήσει, διότι θα είχαμε και αρνητικές επιπτώσεις, τις οποίες κανείς δεν θα ήθελε. Ε, στην Ολομέλεια ίσως θα μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το σημείο περαιτέρω. Και να δούμε ε, τα θετικά ε, των εσόδων από ε, τα στοιχήματα και απευθείας ε, παιχνίδια. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τον πολιτισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την εισηγήτρια για μια πολύ επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς να μιλήσει εκ μέρους του ECR για τους πράσινους. Ναι. Ναι, εν συντομία ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια Πάσχαλ δεν μπορεί να είναι εδώ, είναι ε, ε, Βλέπω ότι υπάρχει κοινή κατανόηση και συνένεση και είμαστε κάπως σκεπτικιστές στο να απαγορευθούν ε, βέβαια υπάρχει πιθανότητα κατάχρησης και πρέπει να το λάβουμε υπόψη αλλά δεν πρέπει να απαγορεύσουμε πλήρως αυτά τα θέματα. Υπάρχει ευαισθησία στο θέμα αυτό και ήταν σημαντικό να αναφέρουμε ότι ε, χρησιμοποιούνται τα έσοδα και για κοινωνικούς σκοπούς που ε, εάν ληφθούν περιοριστικά μέτρα θα έχει επιπτώσεις. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε αφελείς στο τι είναι παράνομος και ποιε είναι οι μορφές, ε, εθιστικές μορφές και θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Αλλά έχουμε πολλά σημεία στα οποία συμφωνούμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια σε αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χοντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και επίσης ε, για τη δουλειά που κάνει και την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζει το θέμα και κοιτώντα και τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τους συναδέλφους όλων των πολιτικών ομάδων οι οποίες ε, στην πλειοψηφία τους με βρίσκουν σύμφωνο διότι είναι σε μια θετική κατεύθυνση αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Θέλω να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι ήδη σε ορισμένες χώρες μεταξύ αυτή και τη δική μου τη χώρα, στην Ελλάδα, στην Τουρκία και σε άλλες χώρες ήδη έχουμε κρίση στο πρόβλημα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου λόγω και στημένων παιχνιδιών. Έχει εμφανιστεί παλαιότερα στην Ιταλία, στη Γερμανία ενδεχομένως και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα είναι ότι πράγματι χρειάζεται ένα πιο ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο. Είναι δύσκολο να το απαγορεύσεις και ο λόγος είναι ότι η δραστηριότητα αναπτύσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, γραφεία στοιχημάτων εδρεύουν κυρίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας όπου γίνονται και στοιχήματα για ευρωπαϊκά αθλητικά γεγονότα, έτσι είναι δύσκολο να το ελέξεις πλήρως. Όμως, συμφωνώ με τους ε, συναδέλφους και με την εισηγήτρια, πρόκειται για μια οικονομική δραστηριότητα η οποία έχει ιδιαίτερη φύση είναι καλό, αλλά δεν πρέπει να υπερβάλλουμε ότι μέσω αυτής της δραστηριότητας ενδεχομένως εξοικονομούνται κονδύλια κυρίως για τον ερασιτεχνικό θα έλεγα αθλητισμό που χρειάζεται μια βοήθεια. Ο επαγγελματικός αθλητισμός έχει τους νόμους τους, έχει τις πηγές τους. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να φεύγει από το μυαλό μας ότι είναι μια δραστηριότητα που καλύπτει, που καλύπτει κρύβει Παράνομε παράνομες δραστηριότητες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καρτέλ και αποτελεί κίνδυνο για τους ανηλίκους. Δεν θέλω να πω περισσότερα παρά μόνο μία πρόταση εκ των τροπολογιών που κατέθεσα λέγοντας ότι και οι άλλες τροπολογίες κατά βάση με βρίσκουν σύμφωνο πρέπει να συζητήσουμε την περίπτωση, να προτείνουμε την περίπτωση της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την ακαιρεότητα και την αντικειμενικότητα του αθλητισμού. Δεν θα λύσει το πρόβλημα αλλά θα έχει μια πιο αυστηρότερη ενδεχομένως παρακολούθηση ίσως εξασφαλιστεί ένα συντονισμένος τρόπος αντιμετώπισης του θέματος καθώς σήμερα με τις εθνικές μόνο προσπάθειες που πρέπει να ενισχυθούν δεν φαίνεται ότι μπορούμε να πάμε σε πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν άλλους τρεις ε, που ανέφεραν ε, ότι έχουν δείξει ότι θέλουν να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Λάγκεν, μετά Σμιτ και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Άλλος παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κονή για την ποιότητα της εργασίας και τις συμβαστικές τροπολογίες που λάβαμε. Εγώ θα ήθελα στις τροπολογίες να επιμείνω σε κάποια σημεία που, σημεία που μου φαίνεται ότι είναι πρωταρχική σημασία. Πρώτα απ' όλα, το γεγονός ότι με τον απευθείας τρόπο ε, που παίζονται τα τυχερά παιχνίδια υπάρχουν περισσότεροι κίνδυνοι από ό,τι όταν παίζει κανείς τον παραδοσιακό τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα, προστατεύσουμε τη ενήλικε, την ακαιρεότητα του αθλητισμού να την προστατεύσουμε. Δεύτερον, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ την απαγόρευση αυτών των παιχνιδιών, τη θέσπιση εθνικού ε, μονοπωλίου και το άνοιγμα τη παραδοσιακή αγορά. Εάν ανοίξει η αγορά, φαίνεται ότι θα ήταν επιθυμητό να μπορέσουμε να εισαγάγουμε ένα σύστημα διοδότησης που να βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες που θα θεσπίσουν οι ενδιαφερόμενοι χωρίς και τα, οι δημόσιες αρχές για να καταπολεμήσουμε Άλλες αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες και τις παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όλα αυτά τα έλαβε υπόψη ε, τα έλαβε υπόψη συμβαστικέ τροπολογίε η συγκεντρία και ελπίζω ότι θα μπορέσουν όταν θα ψηφίσουμε το θέμα τη σήμερα το απόγευμα να επιτύχουμε ευρύτατη συνένεση. Ευχαριστώ. Κύριε Λάγκεν. Ο συνάδελφος ε, από τη Σοσιαλιστική Πολιτική Ομάδα ήδη ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για τις εναλλακτικέ λύσεις ε, μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είτε απαγόρευση δηλαδή είτε κρατικά μονοπόλια. Αυτές ε, είναι οι δύο εναλλακτικέ λύσεις. Όμως επειδή είμαστε στην εποχή του online αυτά δεν γίνονται. Καλύτερα να έχουμε ελεγχόμενες άδειε, ελεγχόμενη αγορά όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μην είναι πλέον παράνομα ε, πολλά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση, σύνδεση online. Εγώ πρέπει να σας πω ότι στη Γερμανία Γερμανία οποιαδήποτε ρύθμιση είχαμε σε σχέση με μονοπόλια και παγορεύσεις δεν λειτουργήσε. Ο μόνον αυτό, αλλά ε, όλοι εκείνοι οι οποίοι ήθελαν και επέμειναν στην ύπαρξή τους κατέφυγαν στην παρανομία. Νομίζω ότι η κυρία Οκονή παρουσίασε μια πολύ καλή γραμμή την οποία πρέπει να ακολουθήσει η γνωμοδότησή μας. Πιστεύω λοιπόν ότι όσον αφορά θέματα καταναλωτών, προστασίας νέων, προστασία του αθλητισμού, παρανομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στην αγορά, ανάμεσα σε όλα αυτά πρέπει να υπάρξει ένα συσχετισμός. Ε, δηλαδή, τα έσοδα τα οποία μέχρι τώρα απέφεραν στο κράτος ε, ήταν χρήσιμα και μειώθηκε και περιορίστηκε η παρανομία. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να στηρίξουμε ένα τέτοιο μοντέλο και όταν μιλάμε, μιλάμε για παράνομα στοιχήματα θα σας πω το εξής, ότι ε, τα παράνομα στοιχήματα δεν φτάνουν ούτε στο ελάχιστο του ύψους των νόμιμων στοιχημάτων. Μιλάμε για νόμιμα στοιχήματα ύψους δισεκατομμυρίων, χωρίς ηθικές αναστολές. Αν λοιπόν ε, πρέπει να απαγορεύσουμε κάτι, τότε θα πρέπει να απαγορεύσουμε κυρίως αυτούς τους ανεύθυνους και όχι γενικότερα το πάθος για στοιχήματα που υπάρχει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ότι εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι ασχολούμαι με τα τυχερά παιχνίδια κάθε εβδομάδα. Από την αρχή με είχε ενθουσιάσει αυτό το θέμα του τυχερού παιχνιδιού. Όμως εγώ δεν ε, παίζω με στοιχήματα απευθείας και άμεσα. Θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στην παράγραφο υπαριθμών 6, για την οποία έχουν κατατεθεί μία σειρά τροπολογιών. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα ε, ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών αν χρησιμοποιεί ή κάνει κατάχρηση αθλητικών γεγονότων σε ολόκληρη την Ευρώπη χωρίς να καταβάλει τίποτα, ένα είδος ας πούμε εισφοράς, ένα είδος τέλους, δεν καταλαβαίνω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Εάν ο τομέας τυχερών παιχνιδιών, ας πούμε, στη Μάλτα, στην Κύπρο, στον τομέα αυτό. Γίνονται στοιχήματα, ας πούμε, για ένα παιχνίδι στη δική μου τη χώρα. Ενδεικτικά το λέω. Αυτά τα στοιχήματα γίνονται online. Είναι προφανές ε, ότι ε, καταβάλλεται ένα τέλος ε, στη δική μου τη χώρα και σε άλλες χώρες αλλά δεν υπάρχει τέλος χρήσης και άδεια για να μπορούν να στοιχηματίσουν για αυτό το παιχνίδι. Συμφωνώ λοιπόν με τον εισηγητή. Είναι αδιανόητον και μάλλον αδύνατον να απαγορέψουμε όλα αυτά. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε αυστηρότερου κανόνε. Δεν ξέρω βέβαια πώ μπορεί να γίνει αυτό, αλλά ίσω ο εισηγητή ε, να έχει κατά νου λιγάκι το πώ μπορεί να λειτουργήσει το θέμα αυτό. Διότι η τεχνική ε, πάντα δυστυχώς προηγείται οι τεχνικοί και οι πονηροί προηγούνται των νομοθετών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ε, πολύ καλή δουλειά που έκανε η κυρία Οκονή και εγώ υπέβαλα κάποιες ε, τροπολογίες και ε, είναι τώρα σε αυτούς τους συμβιβασμούς. Όλα Σμιτ Μα είπε ότι η ακαιρεότητα του αθλητισμού είναι πολύ σημαντική και είναι ένα από αυτά τα θέματα το οποίο αναφέρεται πολύ καλά σε αυτή την έκθεση. Ο αθλητισμός δεν πρέπει να καταντήσει απλά ένα εργαλείο για στοιχήματα και τυχερά παιχνίδια. Έχει τις αξίες του και είναι πολύ σημαντικός. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι ότι τα ατυχήματα, τα τυχερά παιχνίδια δεν είναι οποιαδήποτε ε, επιχείρηση και χρειάζονται περιορισμοί διότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν εργαλεία πρόληψης των καταχρήσεων και να προστατέψουν τους καταναλωτές από, ε, και ειδικά τους ανήλικους ε, και άλλες ε, ευαίσθητες ομάδες που μπορεί να έχουν προβλήματα με το θέμα των τυχερών παιχνιδιών και να κάνουν κατάχρηση. Και επίσης, ε, ο συντονιστικό ρόλος τη Ένωση είναι σημαντικό, διότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο ρύθμισης των τυχερών παιχνιδιών. Για παράδειγμα, αν ένα κράτος-μέλος ε, θέλει να συνεχίσει με το μονοπόλιο, το κρατικό μονοπόλιο, αυτό θα πρέπει να επιτραπεί. Ευχαριστώ. Έχω ένα αίτημα από τον κύριο Σκυλακάκη μπορείτε να προσθέσετε και εσείς το όνομά σας. Ναι, πρώτα θα ε, λάβει το λόγο η ε, ΣΥΡΠΑ και στη συνέχεια εσείς. να πρόβλημα, σας ευχαριστώ. Πρώτα θα ήθελα και εγώ ε, να ευχαριστήσω την Σοφία Κονή για το εξαιρετικό έργο που έχει επιτελέσει την έκθεση αυτή έχει λάβει υπόψη της αρκετές ε, τροπολογίες από αυτές που έχουν προταθεί. Θα ήθελα να τονίσω τρία σημεία στη συζήτησή μας. Πρώτο, λόγω της ειδική φύσεως αυτών των υπηρεσιών αυτού του τομέα ε, των στοιχημάτων όπως και αλκοόλης και του καπνίσματος θα πρέπει να υπάρχει ρύθμιση, ισχυρή ρύθμιση θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες αρχές για τα κράτη-μέλη τι οποίε πρέπει να τηρούν και θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στο θέμα της δομής του μονοπωλίου που πρέπει να είναι καλή γιατί τα έσοδα δεν χρησιμοποιούνται μόνο για τον αθλησμό αλλά και για τον πολιτισμό και για άλλα προγράμματα για την νεολαία. Δεύτερο, χρειαζόμαστε νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, το, το, ε, η μεγαλύτερη απειλή είναι τα διεθνή στοιχήματα σε διεθνές επίπεδο. Ε, και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στην Επιτροπή αυτή για να διασφαλίσουμε ότι και στην Ολομέλεια θα ληφθούν υπόψη σοβαρά αυτά τα σημεία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εντοπίζεται ο παίχτης και εκεί μπορούμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μηχανισμούς εντοπισμού, ε, ταυτοποίησης ε, με ε, την χρήση των ταπεζικών λογαριασμών ή των πιστωτικών καρτών. Και ο παίχτης μπορεί να έχει μόνο ένα λογαριασμό με μια εταιρεία. Διότι αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε να κάνουμε με το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος, ε, και ε, με προβληματικούς παίχτες ε, που έχουν εθισμό στα στοιχήματα. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε την προστασία των παιχτών. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό να τεθεί ένα μέγιστο ποσό απώλειας ζημιάς ανά παίχτη, έτσι ώστε να έχει ένα όριο ο παίχτης και δεν πρέπει να γίνεται ποτέ υπερχρήση και κατάχρηση. Εάν ο παίχτης δώσει αυτό το μέγιστο ποσό σε μια εταιρεία στοιχημάτων θα πρέπει να υποχρεούνται να αποστείλουν αυτές τις πληροφορίες σε όλες τις άλλες, σε όλους φορείς ή τις εταιρείες στοιχημάτων έτσι ώστε να όταν τεθεί το όριο ο παίχτης να μην μπορεί να επερβεί το όριο ε, χρησιμοποιώντας τις άλλες εταιρείες και συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί τα χρήματα. Όταν ε, ε, ανάψει το κόκκινο φως σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Για να είναι αποδοτικό, και εδώ ερχόμαστε στο θέμα της απάτης και του ξεπλήματος και της επιβολής αυτής της νομοθεσίας και των ε, προβλημάτων σε φορολογικά έσοδα. Θα πρέπει να επιμείνουμε στο γεγονός ότι οποιαδήποτε εταιρεία που προσφέρει υπηρεσία στοιχημάτων θα πρέπει να είναι καταχωρημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολύ καλά παραδείγματα αυτών των μηχανισμών. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για τις φορείς πιστοληπτικής ε, ε, ικανότητας των εταιριών και στις παγκόσμιες ε, αγορές δεν μπορεί ε, να ε, μπορούμε να υποχρεώσουμε τις εταιρείε να είναι εγγεγραμμένες και μπορούμε να τις εποπτεύουμε και μπορεί να υπάρχουν προβλήματα επαλήθευσης ε, ειδικά επιγραμμικά online, αλλά δεν είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να δοκιμάσουμε να το κάνουμε και ε, θα υπάρχει συζήτηση για την επαλήθευση των μηχανισμών και επίσης για τα δικαιώματα ε, ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, πρέπει να είναι γεγραμμένες οι εταιρείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, θα πρέπει να υπάρχει η ταυτοποίηση, ο εντοπισμός του παίχτη και τα όρια τα οποία πρέπει να θέτει ο παίχτης. Και το τρίτον είναι η εποπτεία σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει μια αρχή αποπτίας και θα, υπάρχει μια, θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αρχή ε, συνεργασίας ε, της αποπτίας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αποδοτικά τα προβλήματα όταν τα αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, I would also like to thank the rapporteur. Ε, we... Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την συγγήτρια. Ε, γνωρίζουμε ότι τα τυχερά παιχνίδια δεν έχουν σύνορα, δεν γνωρίζουν σύνορα. Υπάρχουν κοινωνικές επιπτώσεις, ε, ε, προκύπτει εθισμός, αναπτύσσονται σχεδόν εγκληματικές ενέργειες. Τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση, αυτό σημαίνει ότι τα κρατικά μονοπόλια δεν αποτελούν πλέον μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη λύση, διότι τα κρατικά μονοπόλια χάνουν τη σημασία τους όταν ε, πλέον ε, τα τυχερά παιχνίδια ε, προσφέρονται όλο και περισσότερο σε απευθεία σύνδεση. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε αυστηρότερους και πανευρωπαϊκούς κανονισμούς για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Στη δική μου τη χώρα, στην Ελλάδα, υπάρχει μια αξιοπερίεργη κατάσταση. Δηλαδή, ιδιωτικοποιήθηκε το κρατικό μονοπόλιο κατά 100%, έχει ιδιωτικοποιηθεί ο φορέας στοιχημάτων μέσα από το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεων και παράλληλα όμως η κυβέρνηση επιθυμεί να δώσει σε αυτό το φορέα παράταση λειτουργίας 10 ετών με τη μορφή μονοπωλίου. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα όσον αφορά τα τυχερά παιχνίδια και νομίζω ότι αυτό το ε, πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουν όλες οι χώρες ε, καθώς επεκτείνεται όλο και περισσότερο το θέμα των ε, τυχερών παιχνιδιών. Κατά την άποψή μου χρειαζόμαστε μια αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική και πρέπει το θέμα του εθισμού να το αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερο συντονισμό. Τα κρατικά μονοπόλια δεν εξέτασαν το θέμα του εθισμού, δεν ασχολήθηκαν καν με αυτό διότι βεβαίως ο εθισμός ε, είναι παντού ίδιος είτε στη Σουηδία είτε στην Ελλάδα. Όσοι είναι εθισμένοι παίκτες ε, τυχερών παιχνιδιών είναι εθισμένοι. Αυτό, ε, από αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε το θέμα και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αναλάβει μία πρωτοβουλία να διατυπώσει προτάσεις πολύ πιο αποτελεσματικά και αποφασιστικά από ό,τι μέχρι τώρα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το όλο θέμα των τυχερών παιχνιδιών στα χέρια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρόεδρος, θα κάνω κι εγώ κάποιες ε, σύντομες ε, παρατηρήσεις ε, απευθύνομαι στην εισηγήτρια. Χαίρομαι πάρα πολύ που εγκρίνατε τις ε, τροπολογίες μου και νομίζω ότι υπάρχουν κάποια θέματα που αφορούν ε, κυρίως ε, στις εγκληματικές δραστηριότητες, στα στημένα παιχνίδια. Υπήρξε τέτοιο θέμα το καλοκαίρι στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Φινλανδία. υπάρχει λοιπόν σαφώς πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι η αγορά online των αθλητικών παιχνιδιών. Μιλάμε για 21,2 δις δολάρια και μιλάμε για μια τεράστια αγορά. Εγκληματικές λοιπόν ενέργειες, ε, στημένα παιχνίδια, αυτά είναι εις βάρος του καταναλωτή τη ε, της οικονομίας, των εσόδων, των κρατικών εσόδων. Άρα δηλαδή ε, πρέπει να αναλάβουμε αυστηρότερες ενέργειες. γνωρίζω ότι ορισμένα κράτη-μέλη ενεχλούνται που η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να αναλάβει περισσότερες ενέργειες για να ρυθμίσει το θέμα. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει υποχρεωτικά ποινικέ ρυθμίσει, αλλά κάτι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Γιατί αλλιώ, αν δεν το κάνουν, θα βλέπουμε όλο και περισσότερα στημένα παιχνίδια στον αθλητισμό. Και αυτό βεβαίω υπονομεύει την ακαιρεότητα του χώρου αυτού. Τέλος, χαίρομαι πάρα πολύ που ε, συμφωνείτε περισσότεροι ότι στον τομέα αυτό πρέπει να στηρίξουν περισσότερο τον αθλητισμό. Όταν μιλάμε για 21,2 δις δολάρια, ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σημαντικό για το κομμάτι που αναλογεί στον αεραστεχνικό αθλητισμό. Από ό,τι κατάλαβα, έχετε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει μελέτε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα και αυτό θα το αναφέρω και στην έκθεση Bowles που και αυτό ασχολείται με το θέμα αυτό ε, για τον αθλητισμό. Ε, και πρέπει να σα πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που εγκρίνεται πολλέ από τι τροπολογίε μα, γιατί πράγματι πρόκειται για ένα τομέα που πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο χώρο για τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Εγώ τελείωσα, θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσά, κυρία Οκονή, ε, και μετά βεβαίω θα λάβει πάλι ε, την Προεδρία η Πρόεδρό μα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπω και ο συνάδελφο Μπαντάρ, χαιρετίζω το γεγονό ότι υπάρχει συνένεση εκ μέρου όλων των πολιτικών ομάδων για το κείμενο αυτό το οποίο κατά την απόψη μου είναι πρωταρχική σημασία. Άκουσα τις παρατηρήσεις σας και συμφωνώ απόλυτα με τις διάφορες παρατηρήσεις που έκαναν οι συνάδελφοι σε σχέση με τα στημένα παιχνίδια, με την παράνομη αγορά, με την προστασία του καταναλωτή, τον εθισμό, τους νέους και τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και την ακεραιότητα του αθλητισμού. Για τον κύριο Ολσμιτ, για την κυρία Μακάρθη, δεν θέλω να πω το εξή. Όσον αφορά τα κέρδη, τα εισοδήματα από τα στοιχήματα και τα τυχερά παιχνίδια online, Είμαι πεπισμένη ότι η ανακατανομή των κερδών αυτών θα πρέπει να ευνοήσει το μαζικό αθλητισμό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Κύριε Οφσμιτ, είπατε ποια είναι η διαδικασία, η μέθοδος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε από νομικής πλευράς την ύπαρξη αυτής της ε, πηγές εισοδήματο Για μένα πρέπει να υπάρχουν από νομικής πλευράς εγγύσεις. Και είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει ποιες είναι οι διαφορετικές μέθοδοι που υπάρχουν ώστε να μπορέσει να επιλέξει την καλύτερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τελικά όσον αφορά τις κυρώσεις, τις παραβάσεις, τα δικήματα. Εγώ, κυρία Πρόεδρε, ήθελα να υπάρξει στην έκθεση αυτή μια κοινό ορισμό και του παραπτώματο και του αδικήματο Ευρωπαϊκού ευρωπαϊκό επίπεδο και των κυρώσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι πρωταρχική σημασία. Και αυτό θα πρέπει να είναι ένας πρώτος αντικειμενικός στόχος της έκθεσής μου, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει στο να έχουμε και πιο φιλόδοξα και συγκεκριμένα κείμενα στο μέλλον για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε σήμερα το πρωί θα ψηφίσουμε και την έκθεση αυτή. Ξέρετε ποιε είναι οι τροπολογίες συμβαστικές. Τώρα περνούμε στο επόμενο θέμα, το σημείο 5. Βλέπω ο Σφέν να τρέχει στη θέση του κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και διατρικέ εταιρείε διαφορετικών κρατών μελών. Συμφώνησα με τον εισηγητή να γίνει και συζήτηση για τα θέματα που εμπεριέχονται στο, στη Λευκή Βίβλο. Πολύ περιορισμένη εμβέλεια για να μπορέσουμε κάποια θέματα από αυτά να τα συζητήσουμε. Δίνω το λόγο στο Σβέν. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, και για το θέμα αυτό είχαμε μια ιδιαίτερα επικοδομητική συνάντηση των σκιωδών εισηγητών η οδηγία περιμητρικής και θηγατρικής εταιρείας μια οδηγία την οποία έχουμε ήδη συζητήσει, αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της κοινή αγοράς. Είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά να μην πλήττονται από τη διπλή φορολόγηση. Παράλληλα βέβαια η απαλλαγή ε, κατά, την, ε, κατά τον επαναπατρισμό των εσόδων ε, μπορεί να ε, καταστεί και αντικείμενο εκμετάλλευση. Γιατί, Γιατί στα διάφορα κρατημέλη υπάρχουν και διαφορετικά συστήματα φορολόγησης. Ο επιχειρηματικός κόσμος ε, μας έχει επισημάνει αρκετές περιπτώσεις ε, αποφυγής διπλής φορολόγησης ή αποφυγής γενικά φορολόγηση. Τελικά τι γίνεται. Οι εταιρείε αυτές δεν φορολογούνται πουθενά και κατόπιν τούτου βλέπουμε ότι η πρακτική αυτή μπορεί να υφίσταται γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ χαμηλή φορολόγηση, χαμηλούς δείκτες φορολόγησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δόθηκε η δυνατότητα να, να ασχοληθούμε με αυτήν την οδηγία και επίσης ε, και να εκφράσουμε την επιθυμία μας ε, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Ε, με λίγα λόγια λοιπόν, η αποφυγή διπλού ε, διπλής φορολόγησης και η πολύ χαμηλή φορολόγηση, αυτά ε, μας δημιουργούν εμάς πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή τα κράτη να ισοσκελίσουν τους ε, προϋπολογισμούς τους. Βλέπουμε ότι υπήρξαν χώρες που το καλοκαίρι αντιμετώπισαν αναταραχές και πάρα πολλοί πολίτες διερωτώνται κατά πόσον είναι σωστό Εν ώψη αυτής της ε, κατάστασης ε, θα πρέπει να δεχόμαστε ότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν φοροφυγάδες, άνθρωποι που μπορούν και πρέπει να πληρώνουν φόρους. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την αναδιατύπωση, εμείς προτείναμε αυτήν την αναδιατύπωση, γιατί αυτό που υπάρχει δεν ταιριάζει ούτε στο πολιτικό ούτε στο οικονομικό σκηνικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ε, συνάντηση ε, των ε, σχεδόν εισηγητών συμφωνήσαμε ότι ε, πρέπει κάτι να κάνουμε για την μη φορολόγηση εταιριών. Να μην ε, μεταφέρουμε το θέμα σε ελληνικές καλένδες, να μην λέμε θα ξεστεί κάπου αλλού και κάποτε, αλλά να επιληφθούμε του θέματος αυτού. Έχουμε λοιπόν τις ε, τροπολογίες που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι στο πλαίσιο της συνάντησης των σχεδόν εισηγητών. Αυτές οι τροπολογίες επί της ουσίας ακολουθούν όλες την ίδια κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω θα τοποθετηθεί εδώ, θα υπάρξει κάποιος εκπρόσωπος Επιτροπής, ε, θα μιλήσω κι εγώ ε, μετά από την παρουσία της Επιτροπής. Εγώ πιστεύω ότι είναι σωστό να γίνει αποδεκτή η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως έχει διατυπωθεί και να μην συνεχιστεί η κατεύθυνση που έχει ήδη χαραχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δέστε παρακαλώ λιγάκι τους προπολογισμού των κυβερνήσεων αυτή τη στιγμή. Νομίζω θα πιστείτε και μόνοι σας ότι υπάρχουν αποχρόντες λόγοι για να ακολουθηθεί μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν που έχετε χαράξει. Ο Ζαν Πολ. Ναι, κάποιες παρατηρήσεις εν συντομία. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπε ο εισηγητής. Θα πρέπει να αποφύγουμε αυτή τη στιγμή να επιμένουμε σε ένα ε, θέμα ανταγωνισμού. Ε, δεν ε, είχαμε, ποια ήταν τα, οι θέσεις των κρατών μελών, κάποιων κρατών μελών που θέλουν να υπάρχει σύγκληση φορολογική που είναι ο πρώτος όρος μια σύγκληση οικονομική. Δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε την οικονομική διακυβέρνηση από μια καλή ε, φορολογική διακυβέρνηση. Δεν πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση σε όλου του κανόνε, αλλά ε, οι κανόνε που παίρνει η Κομισιόν, που προτείνει η Κομισιόν σήμερα και που θα εγκριθούν, θα πρέπει να οδηγήσουν στο αντίθετο αυτό, αυτού που επιθυμούν τα περισσότερα κράτη-μέλη. Δηλαδή, καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση μέσα από αυστηρού φορολογικού κανονισμού και ίση μεταχείριση. Αυτό που προτείνεται ανάμεσα στη Γαλλία και την Γερμανία, εναρμόνιση των φόρων επί των εταίριων και δεν πρέπει να γίνει ε, με φορολογικό dumping ή ε, εξαιρετικό ανταγωνισμό. Σας ευχαριστώ. Ε, Είχα την ευκαιρία να αναφερθώ με τα μου στο γεγονό ότι η Κομισιόν δεν αναφέρθηκε σε ουσιώδη τροποποίηση της ε, αναδιατύπωσης αυτής της οδηγίας και δεν, με αυτόν τον τρόπο δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα του dumping, του φορολογικού και της ε, φοροδιαφυγής. Αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να οδηγήσουν σε αναδιοτύπωση του κειμένου και γι' αυτό η ομάδα μου αποφάσισε μαζί με τον συντάκτη και την Πρόεδρο να χρησιμοποιήσει τον τρόπο χειρισμού με την ε, διοργανωτική συμφωνία για να κάνουμε κάποιες ε, προτάσεις ε, τοπολογιών έτσι ώστε ε, το καθεστώς Μέρφυ να μην οδηγήσει σε μη ε, επιβολή ε, φορολόγησης ή κατώτερη φορολόγηση. Είναι απαραίτητο μια εταιρεία να μην μπορεί να έχει αυτό το πλεονεκτικό καθεστώς μόνο εάν έχει όμως 15% συμμετοχή σε μια εταιρεία σε μια συνεχόμενη διετή περίοδο αυτή η διάταξη θα περιόριζε ε, τα κέρδη. Επίσης, μια μητρική εταιρεία δεν ε, θα πρέπει να μην έχει ε, φόρο επί των κερδών της θηγατρικής, μόνο εάν τα κέρδη αυτά επιβάλλονται στην χώρα της θηγατρικής σε ποσοστό άνω του 15% από το τσιντελιστή που επιβάλλεται σε κράτος μέλος της Ένωσης. Αυτά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι η συγγήτρια για την ομάδα Άλτε. Είναι ένα θέμα το οποίο υποστήριξα ε, στο οποίο υποστήριξα τον εισηγητή, είχαμε, το είχαμε γύρει και στο παρελθόν, πριν από αυτή την πρόταση, το είχαμε γύρει και για την διπλή μη φορολογία με ε, τον Επίτροπο και εν ώψη της ε, ε, οικονομικής κατάστασης που επικρατεί τώρα προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτοί που πρέπει να πληρώνουν φόρουν πληρώνουν φόρουν και υποστηρίζω αυτή την πρόταση λόγω του επίγοντος της κατάστασης και αποφάσισα ως Πρόεδρος να ασκήσω τη διακριτική μου ευκαιρία για να επιτρέψω αυτό το άνοιγμα. Δεν ανοίξαμε όλο την οδηγία, μόνο σε αυτό το περιορισμένο σημείο σχετικά με την διπλή μη φορολόγηση. Με ανησυχεί περισσότερο το θέμα όταν αφορά τη χρήση ε, παραθύρων, όπου τα πλεονεκτήματα των φοροαπαλλαγών που δίδονται σε χρέη φαίνεται να υπερτερούν τον. Ε, εσόδων και τα προβλήματα στα οποία έχουμε επισέλθει αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά, οφείλουν το γεγονό ότι για πολλά χρόνια είχαμε αυτή την πλεονεκτική μεταχείριση ως προς τα χρέη και οτιδήποτε βοηθά στο να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση στο μέλλον θα πρέπει να είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Γι' αυτό ε, αυτό είναι μέρος της μεγαλύτερης εικόνας της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και αυτό ε, θα ε, έλεγα ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να κοιτάξουν τις εισηγήσεις ε, του Κοινοβουλίου με σοβαρότητα και αυτή είναι στιγμή να το κάνουν. Η κρίση και η επίγουσα κατάσταση είναι τώρα και δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αφήσουμε για αργότερα και να δούμε περισσότερες εκθέσεις και να το δούμε στο μέλλον. Είναι θέμα επίγουσας σημασίας. Γι' αυτό υποστηρίζω την κατεύθυνση την οποία έχει ε, πάρει ο συντάκτης, ο εισηγητής. Είναι κανείς που θέλει να λάβει το λόγο. Ναι. Ε, η κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. θα συμφωνούσα ε, με τους προλαλήσαντες. Πρέπει να είμαστε κατά της διπλής φορολόγησης. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε όλες τις πηγές των προβλημάτων στον τομέα ε, φορολόγησης, διότι ε, Έχουμε πολλά και διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Έχουμε πολλές εξαιρέσεις, απαλλαγές και οι εταιρείες ξέρουν πώς να τις αξιοποιήσουν. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε ε, σαφή και διαφανή φορολογικά συστήματα. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο είναι ότι η ουσία οποιασδήποτε δημοκρατικής πολιτικής από την τεμέρη της Βοστόνης είναι η, το, το, το επίπεδο φορολόγησης και ανακατανομής ε, του πλούτου στην κοινωνία. Και πολύ φοβάμαι ότι θέματα όπως το φορολογικό dumping ή ε, υπερβολική, υπερβολικός φορολογικός ανταγωνισμός έρχεται σε αντιπαράθεση με τα φορολογικά συμφέροντα των εθνικών κυβερνήσεων διότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα για τις εθνικές κυβερνήσεις, δηλαδή να είναι ανεξάρτητες στους τομείς αυτούς. Και η υπερκρατική εναρμόνιση μπορεί ε, να θεωρηθεί ως περιττή από αρκετές κυβερνήσεις. Είμαι υπέρ του φορολογικού ανταγωνισμού όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι στην αίθουσα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι Υπουργοί Οικονομικών έχουν τα θέματα τα οποία πρέπει ε, να έχουν τα εισοδήματά τους και τους φόρους που πρέπει να πληρώσουν και πρέπει να δούμε την δομή των φορολογικών συστημάτων. Θα πρέπει να δούμε και τις δύο όψεις του νομίσματος και του προϋπολογισμού. Αυτά ήθελα να πω μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Μεριάν. Ευχαριστώ. Το θέμα ότι θα πρέπει να αντιταχθούμε στις διακρίσεις είναι εμφανές. Θα πρέπει όμως να κοιτάξουμε με ειλικρίνεια και να συνειδητοποιήσουμε ότι η διαφυγή προκύπτει από την νομοθεσία και τότε πρέπει να δούμε ότι η νομοθεσία έχει κάποια ελλείμματα και προβλήματα και θα πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε τα πράγματα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Άκουσα ε, με προσοχή τον εισηγητή που αναφέρθηκε στην πρόταση της Κομισιόν για μια κοινή βάση, φορολογική βάση, ότι θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο την φορολογική βάση αλλά και τους συντελεστές και να συμφωνήσουμε επί των συντελεστών. Θα ήθελα να έχω μια επιφύλαξη εδώ γιατί είχαμε μια ευρεία συζήτηση γι' αυτό στην ομάδα μας. Αυτά είναι πολύ πλατιά θέματα. Αλλά αν υπάρχει αιτιολογική σκέψη, τότε ο εισηγητής ε, θα πρέπει να ε, τα λάβει υπόψη. Υπάρχει διασύνδεση με το CCCTB. Είτε θα έχουμε ένα προαιρετικό σύστημα και η εθνική νομοθεσία θα παραμείνει αναγκαία. Θα πρέπει να έχουμε κατευθυντήρες γραμμές έτσι ώστε να προχωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά όλα αυτά είναι αλληλένδετα θέματα. Και γνωρίζω ότι ο συγγητής ε, μίλησε για το CCCTB, αλλά ε, θα πρέπει να κάνουμε κάτι στο θέμα της ε, αντίθεσης φοροαπαλλαγή. Θα πρέπει το σύστημα του φορολογικού να είναι σαφές και διαφανές και φοβάμαι ότι μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός φορολογικός. Σας ευχαριστώ. Um, ευχαριστώ. Νομίζω ότι η Επιτροπή επιφυλάσσεται. Δεν θα λάβει το λόγο. Τους έχουμε δώσει κάποια μηνύματα. Σβέν, μήπως θέλεις να προσθέσεις κάποια μηνύματα προς την Επιτροπή. Ja, ich ne ich nehme Κοιτάξτε ε, το γεγονός ότι δεν τοποθετούνται ούτε η Κομισιόν ούτε το Συμβούλιο ε, θεωρώ ότι είναι ένα θετικό ε, στοιχείο το καλοκαίρι, οι θερινές διακοπές πολλές φορές ε, ε, ωφελούν στο ότι μπορεί κανείς να προβληματιστεί. Θέλω λοιπόν να πω το εξή ότι όσον αφορά τις ε, τροπολογίες μας, εκεί δεν είναι φιλοσοφική προσέγγιση ε, σχετικά με τα φορολογικά καθεστώτα και τα πλεονεκτήματά τους. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Θεωρώ ότι υπάρχουν, όπως σας είπα, αποχρόντες λόγοι, χώρες ε, που έχουν ε, λίγα δημόσια αγαθά να μπορούν να επιβάλλουν και την ανάλογη φορολογία. Την όλη συζήτηση για τον φορολογικό ανταγωνισμό δεν πρέπει κανείς να την εκμεταλλεύεται έτσι ώστε να ε, υπονομεύονται κάποια θέματα που έχουν σχέση με την εγκατάσταση των εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τι γίνεται, υπάρχουν ε, χώρες ε, με χαμηλότερους φορολογικούς ε, συντελεστές που προσπαθούν να προσελκύσουν ξένες εταιρείε. Νομίζω όμως ότι από αυτού του θέματος και εδώ συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες, κάτι τέτοιο δεν ταυτίζεται με τις ε, αρχές εκείνων ε, που έχουν σκεφτεί το θέμα της αποφυγής του ε, διπλού, της διπλής φορολογίας. Βλέπουμε ότι προκύπτει κατάχρηση όλης αυτής της κατάστασης. Ότι εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί σωστά, είναι σωστή η οδηγία που έχει χαρακτή και γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ που η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα σκεφτούν το θέμα αυτό. Και βεβαίω ε, στη συνάντηση των ε, σκιωδών εισηγητών θα συζητήσουμε τι τροπολογίε με πολύ συναδελφικό πνεύμα και είμαι σίγουρο ότι θα καταλήξουμε σε μια άλλη γραμμή. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ για άλλη μια φορά και την Πρόεδρο και του συναδέλφους και τι συναδέλφου εισηγήτριε που έλαβαν το λόγο σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε μπροστά μας ε, προβλέπει την ψηφοφορία στις 19 Σεπτεμβρίου. Ε, ευχαριστώ λοιπόν πολύ τους ε, συναδέλφους και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης στην αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυρία Λούλιν και η συγγήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την τροποποίηση της οδηγίας της σχετικής ε, για την του κοινωτικού πλησίου πέρσι το να ανοίξει τον Απρίλιο η Επιτροπή. Τι πρότεινα. Να χτενιστεί κατά κάποιο τρόπο το κείμενο που υπήρχε. Δεν πρόκειται για πραγματική επανάσταση. Πρόκειται λοιπόν για μία συζήτηση πάρα πολύ ουσιαστική την οποία θα πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σας κρύβω ότι εγώ ως εισηγήτρια βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Διότι πρόταση με κάνει να έχω κάποια σχόλια αντιφατικά. Κάποτε ήμουν εκπρόσωπος των συμφερόντων και του επαγγελματικού κλάδου και της ε, κοινωνίας γενικότερα που είναι πεπισμένοι για το πόσο σημαντικό είναι το κείμενο αλλά που διαβάζουν με διαφορετικό τρόπο και αντιφατικό αυτά τα οποία περιέχονται στην πρώτη. Με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψη των συναδέλφων για το θέμα αυτό που αφορά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, δεδομένου ότι κατά την άποψή μου και δυστυχώς μόνο στα πλαίσια της διαβούλευσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρουσιάσει ένα ισοσκελισμένο και ε, σωστό κείμενο που να αποτελέσει την βάση επί τη οποία θα λάβει η του Συμβουλίου. Πρέπει να σα πω ότι ακόμη δεν έχω καταλήξει σε συμπεράσματα και βεβαίω θα λάβω υπόψη πάρα πολύ σοβαρά τι απόψει τη πλειοψηφία των συναδέλφων μετά τη συζήτηση που θα έχουμε στην Επιτροπή μας για να μπορέσω να συντάξω την έκθεσή μου. Γι' αυτό θα ήθελα να έχω την υποστήριξη των συναδέλφων για να μπορέσω να υπερασπίσω το αποκλειστικό δικαίωμα και προνόμιο που έχει η Επιτροπή μας για θέματα φορολόγηση. Ορισμένοι από εσά γνωρίζουν κύριε Πρόεδρε ότι η Επιτροπή Ήτρε ζήτησε συνεργασία, ενισχυμένη συνεργασία σε σχέση με την πρόταση οδηγίας αυτή. Τα κείμενα και η πρακτική είναι σαφή. Η φορολόγηση και η φορολογία είναι θέμα αποκλειστική αρμοδιότητα τη επιτροπή μας. Αυτό είναι ένα σύνολο, είναι ένα όλον και δεν μπορούμε ε, να μοιραζόμαστε την Επιτροπή μας σε δέματα φορολόγησης με άλλη Επιτροπή. Δεδομένου ότι το θέμα θα γίνει θέμα που δεν θα μπορούμε, το θέμα αυτό δεν θα μπορούμε πλέον να το διαχειριστούμε, θα είναι πολύπλοκο και το λέγω αυτό λέγοντας συγχρόνως ότι είμαι ανοιχτή σε οποιοδήποτε σχόλιο υποβάλλουν οι συνάδελφοι της Επιτροπής Ενέργειας, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι ότι αυτό το οποίο ήταν αρμοδιότητα κλειδί της δικής μας Επιτροπής πρέπει να παραμείνει ακέραιο. Είναι σημαντικό αυτό, όχι μόνο στα πλαίσια αυτού του φακέλου και επιτρέψτε μου να επιμείνω στο θέμα αυτό. Και βεβαίως αυτό το ανέφερα και στον πρόεδρο της Επιτροπής Ήτρε και ελπίζω, θα το πω μάλλον στον πρόεδρο της Επιτροπής και ελπίζω ότι θα με καταλάβει. Κυρία Πρόεδρε, τώρα θα ήθελα να αναφερθώ γενικά στο περιεχόμενο και στη γενική φιλοσοφία του κειμένου, διότι είναι πρωταρχή σημασία κατά την άποψή μου να γίνει συζήτηση επί αυτού του θέματο πριν να μπορέσουμε να μπούμε σε λεπτομέρειε. Τις λεπτομέρειες που θα μας απασχολήσουν τους επόμενους μήνες για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την φορολόγηση με βέλτιστο τρόπο και να υποστηρίξουμε την αηφόρο ανάπτυξη, όπως λέει η Επιτροπή, προτείνει ο ελάχιστο ποσοστό φορολόγηση να χωριστεί σε δύο μέρη. Πρώτα απ' όλα, ένα μέρος θα αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρωπος που αφορούν τα ενεργειακά προϊόντα που θα καθοριστεί σε 20 ευρώ ανατόνο ε, διοξιδίου του άνθρωπος και ένα άλλο που θα αφορά την, ε, το ενεργειακό περιεχόμενο, δηλαδή την πραγματική ενέργεια την οποία επιτρέπει ένα προϊόντον να μετράτε σε τζουλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αφορά όλα τα καύσιμα και νομίζω ότι η πρόταση αυτή θα βαρύνει πάρα πολύ κάποια ενεργειακά προϊόντα και προβλέπονται βεβαίως και κάποιες περίοδοι μεταβατικοί και περίοδοι προσαρμογής. Χάρη σε μεγάλες περιόδους προσαρμογής για την εναρμόνιση φορολογίας που αφορά το ενεργειακό περιεχόμενο, η Επιτροπή προτείνει αυτές οι περίοδοι να ολοκληρωθούν το, 2023 και να μπορέσουν σε αυτό το νέο φορολογικό καθεστώς να προσαρμοστούν τα διάφορα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά, για μένα εδώ είναι σημαντικό το θέμα της αναλογικότητας. Στο παρόν καθεστώς το ε, ορίζονται τα ελάχιστα κατόφλια και όλα τα κράτη-μέλη βρίσκονται πολύ κάτω από αυτά τα κατόφλια και η αύξηση του κατοφλίου είναι θέμα ε, Αν αλλάξει όμως η μέθοδος και αποφανθούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σέβονται την αναλογία μεταξύ επίπεδου φορολόγησης των διαφόρων ενεργειών που καθορίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή προδιαγραφές και ευρωπαϊκοί κανόνες θα πάρουν άλλη διάσταση, διότι δεν θα πρόκειται πλέον για εφαρμογή του ελάχιστου κατοφλίου, το οποίο είναι κάτι το ξεπερασμένο στα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι θα υπάρξει με απευθείας τρόπο επηρεασμός του πραγματικού επίπεδου φορολόγησης στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πρωταρχική σημασίας και θα ήθελα να ξέρω Εάν οι συνάδελφοι υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση που είναι προφανώς πολύ πιο φιλόδοξη και αποτελεί ένα βήμα προς την φορολογική εναρμόνιση. Θέλουμε αυτή την προσέγγιση όπου τα κράτη-μέλη θα πρέπει αυτή τη στιγμή της οικονομικής κρίσης να φορολογήσουν με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να δοθεί στο ερώτημα αυτό σαφέστατη απάντηση και ελπίζω ότι θα μου τη δώσουν οι συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση προβάλλει άλλα επιχειρήματα τα οποία δεν έχω τον χρόνο να αναπτύξω λεπτομεριακά αλλά αποτελούν ε, πραγματική ενθάρρυνση των ανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ε, των πηγών ενέργειας που ρηπαίνουν λιγότερο. με τη δημιουργία ευρωπαϊκής φορολόγησης και την δημιουργία ε, ίσων κανόνων ανταγωνιστικότητας σε όλη την Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα την μείωση των ε, εκπομπών θερμοκηπίου θα πρέπει να μπορέσουν να συμπληρώσουν το σύστημα εμπορίας μεταξύ των κρατών μελών και θα πρέπει οι τομείς τους οποίους δεν αφορά το σύστημα αυτό να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Δηλαδή, οι μεταφορές, οι μικρές βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις και τα νοικοκυριά. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπόρεσε να φτιάξει ένα πιο συνεκτικό και λογικό σύστημα από το προηγούμενο και αν τα επιχειρήματα υπέρ της καλύτερης χρησιμοποίησης των ενεργειακών πηγών είναι αποδεκτές, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε παρόλα αυτά ότι υπάρχουν επιπτώσεις από αυτή την επαναστατική λύση στη, για την τιμή των ενεργειακών προϊόντων. Πριν να παρουσιαστεί το κείμενο, πρέπει να πω ότι οι διάφορες αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ έντονες. Η εισαγωγή των 20 ευρώ ανατόνο φαίνεται ότι θα αποφέρει 20 δις ευρώ για το σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2020. Εφαρμόζοντας αυτή την ουδέτερη φορολόγηση στην βενζίνη, στο ντίζελ και στα άλλα καύσιμα μετά από μεταβατική περίοδο 10 ετών που θα επιτρέψει στους διάφορες φορείς της αγοράς να μπορέσουν να προσαρμόσουν τις ε, βιομηχανικούς τρόπους παραγωγής τους. Το ντίζελ πρέπει να πω ότι προοδευτικά θα υπαχθεί σε έναν ελάχιστο φόρο αναλύτρο υψηλότερο από αυτός ο οποίος θα επιβληθεί για τη βενζίνη δεδομένου ότι το ενεργειακό του περιεχόμενο ε, είναι διαφορετικό από αυτό της βενζίνης και δεδομένου ότι με το ντίζελ έχουμε περισσότερες εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρωπου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα στη Γερμανία ένα λίτρο ντίζελ κοστίζει 18 cents λιγότερα από ότι ένα λίτρο βενζίνη. Εάν εφαρμοστεί αυτή η φορολογία, το ντίζελ θα κοστίζει 13 του ευρώ περισσότερο από την βενζίνη. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε αύξηση 31 ε, ε, δέκατα ανα λίτρο. Πράγμα το οποίο είναι σημαντικό. Στο θέμα του ντίζελ έχει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι παράλογο ο τομέας της, ε, της αυτοβιομηχανίας να ανησυχεί. Η πολύ σημαντική αύξηση λοιπόν του ντίζελ είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να επομιστούν ούτε οι αυτοκινητιστές που κάθε μέρα πάνε στη δουλειά τους, ούτε η βιομηχανία του κλάδου. Διαρωτώ με λοιπόν και εγώ, όπως και οι συνάδελφοι, αν είναι σωστό αυτό. Παρά το γεγονός ότι δεν συμφωνώ απόλυτα με κάποια ανησυχητικά μηνύματα από την βιομηχανία. Θα πρέπει να πω ότι εάν έχουμε δίζελ πολύ πιο ακριβό από ότι σήμερα θα υπάρξουν προβλήματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το δίζελ είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη. Και καταλαβαίνετε πώς θα επηρεάσει την κατασκευή των οχημάτων η φορολόγηση αυτή στο ντίζελ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει στην Ευρώπη τέτοιου ίδιου ανισορροπία δεδομένου ότι τα διηληστήρια ξέρουμε πώς γίνεται η βενζίνη μετά από εξεργασία τίζελ και λάβετε υπόψη τι ακριβώς γίνεται σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης και τι θα συμβεί για μας με την ε, Ρωσία δίπλα μας. Τα επιχειρήματα λοιπόν αυτά της Επιτροπής θα συνεχίσουν να μας κάνουν εξαρτώμεθα ενεργειακά από το πετρέλαιο σε σχέση με την εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο, το οποίο είναι μια ενεργειακή πηγή η οποία ε, ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο εξαφαλισμένη για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα επιχείρημα θετικό προς το παρόν έχουμε πάρα πολύ λίγα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να αναπτύξει περισσότερο το είδος αυτό της ενέργειας. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά τα διακυβεύματα και τις επιπτώσεις, τις πληθωριστικές που θα μπορούσε να δημιουργήσει η θέσπιση ενός τέτοιου συστήματος. Και νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη η φόβη μας αν λάβουμε υπόψη τη νέα διατύπωση του κειμένου που προβλέπει αυτόματη προσαρμογή πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο νομοθέτης δεν έχει πολύ μεγάλο ρόλο εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να ακούσω τα επιχειρήματα της Επιτροπής η οποία πάντα είναι κατά της αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής των μισθών. Επίσης, λυπούμε διότι δεν αναφέρεται τίποτε για την Ευρωπαϊκή μηχανική Πολιτική στα κείμενα της Επιτροπής και δεν ξέρω αν λαμβάνεται και αυτό υπόψη. Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, ε, ασχολήθηκα και κατά τις διακοπές μου σε μεγάλο βαθμό με το κείμενο αυτό και ξέρω ότι δημιουργήθηκαν και κατά τη μελέτη μου πολλά ερωτηματικά αντί να φωτιστώ περισσότερο για το κείμενο αυτό της Επιτροπής. Περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων και τις υποδείξεις τους ώστε να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε μία γραμμή για το θέμα αυτό φιλόδοξη. Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, αυτά ήθελα να σας πω σε πρώτη φάση και να σας πω και ποιες είναι οι παρατηρήσεις που είχα να κάνω και οι ανησυχίες μου και τα ερωτηματικά μου διαβάζοντας το κείμενο αυτό της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Um, Ευχαριστώ. Ε, μου ζήτησε ο Σκιώδης Τσάλντε να μιλήσει πριν από τους σοσιοδημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και με συγχωρείτε που ζήτησα την άδεια διότι θα πρέπει να πάω στην Επιτροπή Μεταφορών. Η συγγήτρια έχει εισέλθει βέβαια στις λεπτομέρειες ε, της πρότασης που έχει θέσει η Κομισιόν και έχει μιλήσει για τις δυσκολίες που σχετίζονται με αυτό. Βέβαια είναι μια πολύ ε, θετική πρωτοβουλία, αν τη δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προσπαθήσουμε να εσωματίσουμε ένα σύστημα και να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν συγκρίσιμη βάση φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων. Νομίζω είναι θετικό το γεγονός ότι η Κομισιόν έχει προτείνει αυτή την πρόταση. Είναι μια θαραλέα πρωτοβολία, γιατί όπως είπε και η συγγήτρια, με Υπάρχουν ε, πολλές πολιτικές που ε, εμπλέκονται και πολλά, ε, πολλές σοβαρές πολιτικές διακλαδώσεις όταν μιλάμε για αύξηση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων. Είναι κάτι που θα είναι αναπόφευκτο στο μέλλον. Στο δικό μου κρατός μέλος, για να αναφερθώ μόνο σε ένα, οι φόροι επηρεάζουν μεν ε, τον καθορισμό των τιμών. Εδώ θα πρέπει να δούμε χαμηλότερη κατανάλωση δίζελ, αλλά οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας το βλέπουν ως ένα μεγάλο μέρος της μείωσης ε, των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακο που σχετίζεται με την τεχνολογία δίζελ. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα συμβάσουμε αυτό με την πρόταση. Θα πρέπει να εξετάσουμε από πολύ κοντά το κείμενο ε, και τα επόμενα χρόνια θα είναι σημαντικό. Είναι μια μεταβατική φάση προς το μέλλον. Τα επόμενα μερικά χρόνια θα πρέπει ε, τα κέρδη μας ε, σε ό,τι αφορά τις μειώσεις διοξιδίου άνθρωπου να γίνουν στην τεχνολογία του ντίζελ. Στη χώρα μου υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν αγοράσει ντίζελοκινητήρες γιατί είναι πολύ πιο φτηνό το ντίζελ από την βενζίνη. Βλέπουμε ότι το 3 τέταρτα των αυτοκινήτων που κινούνται με ντίζελ ε, πολλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει να έχουμε αυτό ε, το παράγοντα κατά νου. Τώρα, αν μιλάμε για την χρήση ντίζελ για επαγγελματικά οχήματα, Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον δίζελ και την βενζίνη για πολλές ε, ε, εταιρείες μεταφορών και είναι πολύ σημαντικό για αυτές τις εταιρείες. Θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τι είναι εφικτό και τι δεν είναι. Επιπρόσθετα τώρα. Βλέπουμε τον ε, φόρο των καυσίμων ταυτόχρονα δεν υπάρχει ισοσκέλεια ανάμεσα στην χρήση των μορφών ε, συγκοινωνίας. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια. Αν ε, μιλάμε για ίση μεταχείριση ανάμεσα στα διάφορα μέσα ε, συγκοινωνίας, θα πρέπει επίσης να μην έχουμε και υπερβολικά αρνητικό αντίκτυπο για ορισμένα θέματα που χρειαζόμαστε στην για να συνεχίσει να κινείται η οικονομία. Τώρα, στο Κοινοβούλιο ε, μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε. Η Επιτροπή μας ε, μπορεί να το κάνει, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε η Επιτροπή που θα συνεχίσει να ε, συντάσει αυτή την έκθεση. Δεν πρέπει να επαναχωρήσουμε στο μέτωπο αυτό. Αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι όμως τώρα, θα πρέπει να έχουμε ευρεία πλειοψηφία υπέρ της γνωμοδότησης ε, την οποία εμείς εκδίδουμε ως Κοινοβούλιο, διότι αλλιώς δεν θα μας εισακούσουν. Ε, τώρα, προσβλέπω στη συζήτηση στο Συμβούλιο, θα είναι μία από τις πιο συναρπαστικές συζητήσεις που θα ανέμενε κανείς στους επόμενους μήνες. Αλλά είναι ενδιαφέρουσα η αρχή, το γεγονός ότι δεν μιλάμε για κατανάλωση, όταν μιλάμε για την ελάχιστη φορολόγηση, τον ελάχιστο φόρο ε, αλλά μιλάμε για το ε, περιεχόμενο ε, εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα. Ε, καταρχήν, αυτή είναι πολύ θετική ιδέα. Δεν πρέπει να απομακρυνθούμε πολύ από αυτή την αρχή. Θα πρέπει να δούμε την μεταβατική περίοδο, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ε, να δούμε ποιες θα είναι οι μεταβατικές περιόδοι που θα απαιτηθούν στις διάφορους κλάδους της ε, βιομηχανίας και που θα επηρεαστούν. Θα πρέπει επίσης να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της επικουρικότητας. Πώς θα επηρεάσει αυτό το σύστημα το φορολογικό ε, στα προϊόντα ενέργειας και με σε ποιο βαθμό θα περιορίζεται η ελευθερία των κρατών μελών. Αν ε, μιλάμε για ελάχιστο συντελεστή, θα πρέπει να δούμε και τα μελλοντικά στάδια. Θα ήταν πρόωρο να λάβουμε κάποια θέση εδώ, αλλά ε, θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθούμε στα σημαντικά θέματα πρώτα. Άρα, κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι περνούμε πολύ ενδιαφέρον ε, μια ενδιαφέρουσα φάση στο θέμα αυτό με πολιτικές επιπτώσεις. Είπα ότι ε, πίστευα ότι η πρόταση της Κομισιός Κομισιόν ήταν λογική και πήρα πολλά emails από ε, διάφορους οργισμένους που μου λένε πρώτα με ενθαρρύνεται να αγοράζω διζελοκινητήρες και μετά ανεβάζετε τους φόρους στα δίζελ. Ε, υπάρχουν πολλά συναισθήματα και δεν είναι πάντα λογικά. Ε, κυρία Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω ελεύθερα στο θέμα αυτό, διότι είναι η τελευταία φορά που παρευρίσκομαι εδώ σε αυτήν την Επιτροπή, διότι από την επόμενη εβδομάδα ε, και ο Φιλίπ θα με διαδεχθεί. Θα ακολουθήσει ε, το έργο αυτό με ε, τον ίδιο ενθουσιασμό. Ευχαριστώ τους συνελεύθερους για την συνεργασία που είχαμε μαζί. Δεν ε, θα έχω πια τις επιπτώσεις των λόγων σε αυτές τις συζητήσεις. Σας εύχομαι επικοδομητική συνέχεια στη συζήτηση. Ευχαριστώ, Ντέρκ. σας εύχομαι το καλύτερο στα χρόνια της σύνταξης. Ε, θα επανέλθουμε τώρα στον Όλεκ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Κομισιόν έχει κάνει τη δουλειά της. Θα πρέπει να δούμε την πρόταση και να δούμε ότι είναι ισορροπημένη. Υπάρχουν όμως κάποιες αδυνάμεις, κάποια προβλήματα για Γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε από κοντά. Αλλά η αρχή στην οποία στηρίζεται είναι καλή και γερή. Ιδιαίτερα όταν η Κομισιόν πρότεινε ε, ότι ε, ε, αυτό εδώ μιλάμε για την μείωση των εκπομπών και για τις ΑΠΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα και υπάρχει μια θετική κατεύθυνση στο σύστημα εμπορίας ε, ε, εκπομπών. Ο εξυγχρονισμός αυτό είναι σαφές. Ε, η Κομισιόν έχει φέρει καλές λύσεις σε προβλήματα. Τώρα, αν δούμε την ενεργειακή φορολόγηση και την οδηγία ε, είναι ένα εργαλείο επιτάχυσης ε, της διαδικασίας. Ε, περνάμε την φορολόγηση σε ένα άλλο παραγόντο, την ενέργεια, και αυτό θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα, θα βελτιώσει το περιβάλλον χωρίς να υποβαθμίσει το περιβάλλον. Πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει βέβαια να την επεξεργαστούμε για να δούμε την ανταγωνιστικότητα των εταιριών. Ε, γενικά, νομίζω η πρόθεση της ε, πρότασης αυτής είναι καλή. Εδώ βέβαια δεν ε, είμαστε πρώτοι στην πράσινη τεχνολογία. Υπάρχει ανταγωνισμός που είναι όλο ένα πιο δύσκολο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά αν δούμε το εισαγωγικό μέρος, την εισαγωγική φάση, θα υπάρξουν θα υπάρξει κάποια αντίθεση στην, γενικά και σε, σε ειδικά σημεία της πρότασης, αλλά υπάρχει ένας άλλος τομέας που στηρίζεται σε πιο γενικά επιχειρήματα, ότι στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξουμε φιλόδοξη σε ε, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τομέα του περιβάλλοντος και της εσωτερική αγοράς. Θα πρέπει να δούμε την Ευρώπη ως σύνολο. Το Συμβούλιο δεν θα ε, είναι πολύ ε, ευτυχές σε αυτό το θέμα. Τώρα στα ελλείμματα και στα προβλήματα. Θα πρέπει να τα αναλύσουμε και να τα δούμε λεπτομερώς. Στην πρόταση εδώ. Θα είναι δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο να προσπαθήσουμε να δούμε μια σφαιρική λύση, γενική λύση, ακόμη και τώρα. Εάν μιλάμε για ε, συμφωνία επί των λεπτομεριών, η Επιτροπή θα πρέπει να υλοποιήσει αυτές τις προτάσεις στη λεπτομέρεια. Αλλά θα πρέπει ίσως να αφαιρέσουμε την φορολόγηση στην διεθνή αεροπορία και στον τομέα των ναυτιλιακό. Ε, βλέπουμε κάποιες οδηγίες. Δεν νομίζω να υπάρχουν σοβαρές αλλαγές βραχυπρόθεσμα, αλλά ε, κινούμε προς την σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τα οχήματα. Δουλεύουμε πολύ σκληρά να βρούμε καλές λύσεις ε, ανάμεσα στη χρήση του ντίζελ και της βενζίνης. Και πάλι η αρχή της φορολόγησης θα έχει επιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια όταν μιλάμε για τη φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, όταν μιλάμε για ευρυδικά οχήματα. Θα πρέπει να ε, δούμε την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας και της χρήσης της στον τομέα των οχημάτων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, αυτά τα προβλήματα, να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες που έχουν ήδη υψηλά ενεργειακά κόστη, ε, και, ε, αλλά πρέπει να, είναι, ε, να διασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση είναι επικερδείς. Τώρα, αν δούμε τους μηχανισμούς καθορισμού των τιμών, ε, υπάρχει απαλλαγή από σε κάποιους τομείς θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε τους ελάχιστους ε, φορολογικούς συντελεστές. Ε, θα πρέπει να δούμε προσαρμογές στις τιμές ε, του συστήματος εμπαρίας εκπομπών. Και πάλι εδώ βλέπουμε το θέμα του φορούνται de Είναι κάποιες από τις προκαταρκτικές μου απόψεις αυτές και βέβαια προσβλέπω σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Ευχαριστώ την κυρία Λούλιν για την πολύ περιεκτική δουλειά που έκανε και για την παρουσίασή της και λυπάμαι που έπρεπε να αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών για να ασχοληθεί με αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το μέρος του ECR. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να υπογραμμίσω ότι προφανώς επιθυμώ και επιδιώκω τη συνεργασία με την γοητευτική κυρία Λούλινγκ. Πέρα από αυτό όμως θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα που ετέθησαν κατά τη διάρκεια της ε, συζήτησης. Πρώτα απ' όλα, ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λούλινγκ, για την θαυμάσια εισήγησή σας και ε, για τον αρκτήριο λάκτισμα που δώσατε στη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω τουλάχιστον τέσσερα σημεία που με απασχολούν. Ε, το πρώτο θέμα, το οποίο ευτυχώς ή δυστυχώς ε, για ορισμένους από εσάς, ε, είναι κατά την άποψή μου καθοριστικής σημασίας. Πρόκειται για την τιμή της ενέργειας. Όπως και στην περίπτωση άλλων τιμών, είναι συνάρτηση προσφοράς και ζήτησης. Και κάθε προσπάθεια να επηρεάσει κανείς τιμές. Με τεχνητό τρόπο κάθε τέτοια προσπάθεια είναι επιζήμια ε, για το σύνολο της αγοράς. Αυτό είναι το πρώτο που με απασχολεί. Το δεύτερο είναι το εξής ε, έχει σχέση με τους ε, καταναλωτές. Κατά την άποψή μου, ο καταναλωτής είναι καθοριστικός παράγων στην αγορά όχι τόσο ο νομοθέτης. Ο καταναλωτής ε, και η συμπεριφορά του είναι καθοριστική σημασίας. Είναι ε, προφανές ε, ότι οι καταναλωτές έχουν τις δικές τους προτιμήσεις για τα αυτοκίνητά τους, για το τι καταναλώνουν. Και ως εκ τούτου η συμπεριφορά τους μπορεί ε, να είναι μειονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι που ορισμένοι από εσά ε, ήδη αναφέρετε. Ε, πρόκειται για τις κοινωνικές συνέπειες. Οι κοινωνικές συνέπειες από την αύξηση της άμεσης φορολογίας. Μπορώ να σας πω, να σας παραπέμψω στο παράδειγμα της Τσεχίας. Η ηλιακή ενέργεια και η ευρεία κατανάλωσή της τελικά οδήγησε σε αύξηση ε, για τον καταναλωτή της τάξης του 10% στην ενέργεια, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και το τέταρτο που θέλω να επισημάνω είναι η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, μέσα στο παγκόσμιο αυτό σκηνικό που υπάρχει. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, να επιδιώξουμε το καλύτερο, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτύσσεται σε ένα διεθνές πλαίσιο, πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου, και καταλήγοντας, να πω και πάλι, προσβλέπω στη συνεργασία με την κυρία Λούλινγκ, η οποία είναι μια πολύ λογική και ευαίσθητη συνάδελφος. Εκ μέρους των Πρασίνων, ο Φιλίπ. ο Φιλίπ ε, έπρεπε να ψηφίσει στην Ήτρε ε, και ακόμα δεν έχει συνέλθει. Μερικέ φορέ εκεί οι ψηφοφορίε είναι πολύ δύσκολε Να πω λοιπόν το εξή εγώ. Ε, θα σχολιάσω ορισμένα από αυτά που ελέγχθησαν. Καταρχήν, συμφωνούμε με την ε, γενικότερη άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής επί του θέματος. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι εμεί, επειδή είμαστε Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, πρέπει να εξετάσουμε λίγο το στοιχείο του, το, το οικονομικό μέγεθο, την οικονομική διάσταση που διαμορφώνει τις τιμές. Ο συνάδελφος από την Τσεχία ε, παρέπεμψε στην ε, αποτελεσματικότητα των αγορών ε, και τα κράτη πρέπει να έχουν το όπλο της φορολογίας για να επεμβαίνουν ε, στο μηχανισμό καθορισμού τιμών αλλά και σε νεοκλασικές οικονομίες υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις ε, ε, στην αγορά. Δηλαδή παραγωγή καταρχήν πετρελαίου, παραγωγή αερίου, συμπαραγωγή, πού παράγονται όλα αυτά, αυτό επηρεάζει. Μετά κλιματολογικές συνθήκες, ε, οι μελλοντικές ε, γενιές ε, που θα είναι σε πολύ χειρότερη θέση από εμάς θα κληθούν να καταβάλουν πολύ μεγάλη τιμή για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να διορθώσουμε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις οι εξωτερικοί αρνητικοί παράγοντες δεν συμπεριλαμβάνουν του υπολογισμού ε, και απλά μόνο υπολογίζονται στη φορολογία. Η Κομισιόν λέει ότι μάλλον με την παρέμβασή της τώρα οι αγορές ε, καθορίζουν καλύτερες, πιο σωστές τιμές. Αυτό ε, το είπε και ο Νίκολα Στέρν, ο οποίος στην οικονομική κοινότητα έτυχε μεγάλης υποστήριξης πέρα από τη συνήθη μόχλευση που εφαρμόζεται. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει τρόπους για να λειτουργεί καλύτερα το σύστημα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να διαπιστώσει κανείς ότι οι διαφορές στη φορολογία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή οδηγούν σε παράλογες συμπεριφορές. Λόγω λοιπόν του ότι υπάρχουν διαφορές στα εθνικά συστήματα φορολογίας για το θέμα της ενέργειας έχουμε ε, χρήστες ε, που χρησιμοποιούν ακόμα και πιο ρηπογόνες μορφές ε, κατανάλωσης που δεν θα το έκαναν αν τελικά τα συστήματα ήταν περισσότερο εναρμονισμένα. Άρα πρέπει να υπάρχει κοινή αγορά. Ε, καμία συζήτηση από αυτού. Κατόπιν, οι εμπειρογνώμες κομισιών για κλιματολογικά θέματα, αλλά και πολλοί άλλοι επιστημονικοί παρατηρητές προτείνουν ότι για να υπάρξει κάποια διαφορά σε επίπεδο κλίματος σε σχέση με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι 30 αλλά 20 ευρώ για κάθε τόνο ε, εκπομπής ε, διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό ίσως είναι πιο λογικό ε, και σε σχέση με μακρόπνοες προοπτικές. Αν όμως επιτύχουμε την εναρμόνιση και ε, απομακρύνουμε κάποια αρνητικά κίνητρα, ενδέχεται σε κάποιους τομείς να υπάρξουν ανατιμολογήσεις. Αυτές λοιπόν οι αυξήσεις τιμών ενδέχεται να έχουν κάποιες συνέπειες. Ε, κατόπιν τούτου ε, επισημαίνονται οι κοινωνικές συνέπειες και συμφωνώ ότι οι κοινωνικές συνέπειες της φορολογίας από τη φορολογία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υπάρχουν κάποιες διορθώσεις ε, στις, ε, στην χρήση των κονδυλίων. Τα κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιούνται για να μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ε, να μειώνεται, να μειωθεί η φορολογία ε, της εργασίας, κυρίως για τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Άρα δηλαδή δεν είναι απαραίτητα αρνητικές επιπτώσεις ε, από την ε, κλιματολογική φορολογία όπως θα τη χαρακτηρίσω. Και τέλος, στην πρόταση της Κομισιόν δεν είναι σωστό να, λένε, να αναφέρεται ότι εξαιρούνται τα καύσιμα της αεροπλοείας. Αυτή είναι μέρος του ε, προβλήματος. Είναι η σημαντικότερη πηγή εκπομπής διοξιδίων του άνθρακα στον τομέα των μεταφορών. Ε, και όπως επισήμανε και η συγγήτρια, υπάρχει και μία άλλη μορφή αρνητικών κινήτρων ε, όσον αφορά τα διάφορα μέσα μεταφοράς. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το θέμα αυτό και πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή το θέμα επήγει για οικονομικούς λόγους, για κλιματολογικούς. Αν τα φορολογικά κίνητρα δώσουν το σωστό μήνυμα, δηλαδή να προχωρήσουμε πιο γρήγορα σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας, τότε αυτό ε, θα είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και για την ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία. Το γεγονός ότι υπάρχει όμως στεναρή αντίδραση σε αυτό που σου λέω, αυτό δεν ωφελεί μακροπρόθεσμα τον τομέα. Γι' αυτό πρέπει να στηρίξουμε την Επιτροπή στο να υπάρχουν ταχύτερες εξελίξεις γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να δούμε ε, αυτοκίνητα από την Κίνα που θα έχουν κάνει εκείνα το πρώτο βήμα και θα ε, δούμε επίσης βιομηχανίες να εγκαταλείπουν την Ευρώπη. Απλά και μόνο γιατί επιμένουμε στη διατήρηση κεκτημένων του παρελθόντος. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν πολύ πιο σωστό να προχωρήσουμε ταχύτερα, πολύ πιο σωστό από το να περιμένουμε να υπερισχύσουν στην αγορά άλλοι παράγοντες. Συνάδελφος Πόρτας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλές Σωστές παρατηρήσεις έγιναν κατά την άποψή μου. Συμφωνώ με τους γενικούς στόχους που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για την φορολόγηση ως μέσον πολιτικής και ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Ξεκινώ από μια διαπίστωση που έκανε ο συνέλφο Τέρξ και με την οποία συμφωνώ. Και όπως είπε και η συγγήτρια, οι προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν επανάσταση για τις τιμές της ενεργειακές. Επανάσταση γιατί, διότι γενικά προβλέπει αύξηση των τιμών. Μπορούμε να φανταστούμε μία ουδέτερη φορολογική πολιτική όσον αφορά την τιμή. Αλλά είναι νομίζω λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές αυτές κατευθυντήριες γραμμές να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Εγώ θα ήθελα να τονίσω τρία θέματα τα οποία κατά την άποψή μου είναι πρωταρχική σημασία από κοινωνική άποψη. Κυρίως για τις ε, κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των προτάσεων όσον αφορά τους συμπολίτες μας. Πρώτα απ' όλα, είμαι υπέρ όλων όσων λέγονται υπέρ το ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να επωφελούνται από ευελιξία για να εφαρμόζουν αυξήσεις ή μειώσεις για τα νοικοκυριά που έχουν τις περισσότερες οικονομικές δυσκολίες. Γι' αυτό για μένα είναι πρωταρχή σημασία στα πλαίσια της επανάστασης αυτής για τις τιμές. Το είδος χρησιμοποίησης της ενέργειας και ο αποδέκτης της θα πρέπει να είναι σημαντικές στον καθορισμό της φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων. Διότι υπάρχει υποχρεωτική κατανάλωση, αμφιλεγόμενη και κατανάλωση η οποία δεν είναι καθόλου απαραίτητη. Είναι επιφανειακή. Και αυτού του είδους η κατανάλωση η τελευταία θα πρέπει να πληρώνει. Δεύτερον, μία ιδέα η οποία θα συζητηθεί στο επόμενο θέμα, η ιδέα του Φιλίπ Λαμπέρ, για να δούμε αν θα επιβάλλουμε πράσινο ΦΠΑ στον ενεργειακό τομέα. Αυτού του είδους το μέσον μπορεί να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό για τον προσανατολισμό που θα δώσουμε στη βιομηχανική μας πολιτική. Τρίτη παρατήρηση. Έχω μια αμφιβολία η ιδέα να μην κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ του εμπορικού δίζελ και του, του, για εμπορικούς λόγους και μη κατά την άποψή μου μπορεί να είναι σωστό θεωριστικά αλλά πιστεύω ότι στην πράξη είναι δύσκολο αν δεν υπάρξει μία μεγάλη μεταβατική περίοδος να δούμε τι ακριβώς επιβάλλεται στις ε, ε, μεταφορές με ιδιωτικά αυτοκίνητα σχέση με τη μεταφορά ε, των μέσων κοινή μεταφοράς. Και εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί διότι τα δημόσια μέσα μεταφοράς θα πρέπει να τα υποστηρίζουν. Τώρα, σε σχέση με τα βιοκαύσιμα που προτείνει η Επιτροπή. Έχω ένα ερωτηματικό και αυτό είναι θέμα συζήτηση συζήτησε μία επόμενη φορά. Η γενικότερη τάση είναι όντως να ευνοήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά βλέπω ότι υπάρχει εδώ και το θέμα της πυρηνικής ενέργειας και τι χρήση θέλουμε να κάνουμε. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ευχαριστώ. Τελείωσαν οι σκιώδεις ηγητές, δεν έχω άλλο συνάδελφο που ζητήσει το λόγο. Έχουμε αρκετό χρόνο στην διάθεσή μα Αστρίντ. Θέλει να πεις κάτι τελειώνοντα. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδες ηγητές. Ω, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Η Κομισιόν, θέλουμε να ακούσουμε, θέλετε να ακούσετε και την Κομισιόν. Πολύ σύντομα θα δώσω το λόγο και στην Κομισιόν. Νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει αν θέλει οπωσδήποτε η Κομισιόν να πει κάτι, της δίνει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Λούλιν για την ε, ανοιχτή και επικοδομητική εισαγωγή της σε σχέση με την πρόταση αυτή. Βεβαίως, βλέπουμε με ικανοποίηση ότι αναγνωρίζεται ότι είναι πιο λογική και πιο ε, συνεκτική η πρότασή μας και περιέχει κάποιες θετικές παρατηρήσεις. Πράγμα το οποίο ανέφερε ο της και ο κύριος Στέρκ. Όντως, έχετε επιτάπητος μία μεγάλη αλλαγή δεδομένου το θέμα της ενεργικής φορολόγησης σήμερα δεν, είναι ένα, δεν βασίζεται σε ένα βιώσιμο σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει. Όπως αναφέρθηκε και από πολλούς συναδέλφους σας, τα βασικά ερωτήματα είναι, είναι σωστό η, να πληρώνει ο άνθρακας που είναι το πιο ε, το καύσιμο το οποίο ρηπαίνει περισσότερο μικρότερο φόρο θα είναι σωστό να υπάρχει τέτοια αύξηση στον διζελ μετά από την φορολόγηση αναφέρθηκε για αυτό το θέμα και το βιοντίζελ, τα βιοκαύσιμα θα πρέπει να έχουν την ε, ίδια μεταχείριση ενώ πραγματικά ρηπαίνουν λιγότερο. Τα κρατημέλη με την στρατηγική του 2020 ε, πραγματικά έχουν δώσει απάντηση, διότι είπαμε για το 2020 θέλουμε να έχουμε ε, λιγότερο κατά 20% κα, ε, ε, καύσιμα που ρηπαίνουν, 6,5% Αυτό είναι κάτι το οποίο εξηγείται στις ε, διάφορες προτάσεις και ξέρουμε ότι υπάρχουν παρόλα αυτά, δεν υπάρχει γενική συμφωνία, υπάρχουν διάφορες ανησυχίες οι οποίες είναι λογικές και εκφράζονται από την βιομηχανία και γι' αυτό προβλέπονται μεγάλες μεταβατικές περίοδοι και αυτό εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι για πρώτη φορά υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ ε, του συστήματος εμπορίας των ρήπων και των ενεργειακών προϊόντων. Όσον αφορά την ε, τεχνολογία και τη μηχανία που αφορά την αυτοκίνητοβιομηχανία και τον ντίζελ. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι ένα συνεκτικό κείμενο. Υπάρχει ε, τα, πλεονεκτήματα από τη χρησιμοποίηση κινητήρων δίζελ σε σχέση με τους κινητήρες βενζίνη δεν επηρεάζονται από αυτή την πρόταση και βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί η ζήτηση σε αυτοκίνητα με κινητήρα δίζελ. Δεδομένου ότι αυτά του είδους τα οχήματα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Δεν θα υπάρχει επίσης συστηματική επίπτωση για στην ε, πληθωρισμό για δύο λόγους, διότι τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να μπορούν να επιβάλλουν τους φόρους που επιθυμούν και να μπορούν να αναθεωρούν τα συστήματα φορολόγησης βάσει των δικών τους ε, αναγκών και τα θέμα των ε, κατοφλίων και η επιβολή των εμέσων φόρων είναι ένα σύστημα το οποίο θα ομαλοποιηθεί. Λαμβάνεται επίσης ε, υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούν χωρίς να υπάρχει μεταβατική φάση αλλά σε μόνιμη φάση να εξαιρούν πλήρως ε, τα καύσιμα για θέρμανση των οικοκυριών εάν θεωρούν ότι αυτό είναι η καλύτερη λύση. Βεβαίω ε, μπορούμε να συνεχίσουμε και με το εμπορικό δίζελ και πάρα πολλά άλλα παρεμφερή αλλά εγώ δέχομαι αυτό που μου είπατε ότι ε, είναι πολύ χρόνο. είμαστε υποποίηση χρόνου. Σταματάω λοιπόν εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, για τις επικοδομητικές του παρεμβάσεις και προσβλέπουμε στην τελική διατύπωση του θέματο. Τώρα η Άστριτ μπορεί και πάλι να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε γιατί δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους γιώδεις εισηγητές. Πιστεύω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η θέση του καθενός. Τους ευχαριστώ κυρίως για τις προτάσεις και για την πολύ σαφή τους τοποθέτηση όσον αφορά τις μεγάλες προκλήσεις. Προτείνω να οργανώσουμε όχι μια κρόαση γιατί είναι πολύπλοκο αλλά ένα σεμινάριο αν θέλετε με εμπειρογνώμονες. Μιλήσαμε για αυτό το θέμα με την ε, γραμματεία. Ίσως στις 5 Οκτωβρίου θα μπορούσαμε να το οργανώσουμε γιατί εγώ θα ήθελα οι εμπειρογνώμονες να μπορέσουν να μας εξηγήσουν ποιες είναι οι δικές τους απόψεις και οι δικές τους ανησυχίες. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ενδιαφέρον για όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Και θα ήθελα να πω ότι μπορώ να έρθω αμέσως σε επαφή και με τους κοιόδης εισηγητές. Θα προσπαθήσω να τους συναντήσω, να συζητήσουμε το όλο θέμα, διότι όπως βλέπετε το πρόβλημα είναι πάρα πάρα πολύ αντιφατικό και περίπλοκο. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, εγώ θα ήθελα να κάνω ό,τι έκανε και το Συμβούλιο και μου είπαν δεν έκανε τίποτε. Οι Πολωνοί δηλαδή, αν είμαι καλά πληροφορημένοι, δεν προτίθενται να δώσουν προτεραιότητα στο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, από μεριάς Συμβουλίου, ξέρουμε βεβαίως ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλήσεις απόψεων, αλλά γνωρίζουμε ότι η Πολωνική Προεδρία δεν προτίθεται να επιταχύνει τα πράγματα ούτε καν αν κατάλαβα καλά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη. Και εμείς πριν να ορίσουμε τις δικές μας προθεσμίες θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους επίσης για την θέση μας σε σχέση με την Επιτροπή Ήτρε. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να δώσει να καταλάβει η ΤΡΕ ότι επιμένουμε στη θέση την οποία εκφράσαμε και γραπτός. Αυτό θα ήθελα να πω κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να οργανώσουμε αυτό το σεμινάριο, αυτό το workshop το συντομότερο δυνατό, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε και τους ενδιαφερόμενους που θα μπουν σε λεπτομέρειες και τους μεν και τους δε, διότι Πιστεύω ότι αυτό θα μας βοηθήσει όλους. Γι' αυτό θα πρέπει να καθορίσουμε τις ε, προθεσμίες και τις ημερομηνίε των εργασιών μας σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζουμε όσον αφορά την, σχέση, την ε, ε, θέση που θα διαμορφώσει το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ε, προφανώς ε, είμαστε από ό,τι φαίνεται η πλέον δημοφιλής επιτροπή στο Κοινοβούλιο γιατί από ό,τι φαίνεται όλες οι άλλες επιτροπές θέλουν να μοιραστούν ε, πράγματα με μας. Και επειδή αναφέρεται η ενέργεια, παρότι έχει σχέση με τη φορολογία, το θέμα υποτίθεται ότι υπάρχει της αρμόδιας επιτροπής ΙΤΡΕ. Ίσως θα πρέπει να το θίξω το θέμα αυτό στη διάσκεψη των Πρόεδρων, αλλά από ό,τι φαίνεται όλα τα θέματα ε, κατά κάποιον τρόπο μπαίνουν και στις δικές μας αρμοδιότητες. Και εδώ θα με στηρίξει φαντάζομαι η Άστριτ όταν μας δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουμε την άποψή μας δεν θα πρέπει βέβαια να ε, αποποιούμεθα αυτού του δικαιώματο. Ελπίζω, με πάση περιπτώσει, αυτή τη φορά να μην χρειαστεί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να βρεθεί μια τελική λύση. Το σχέδιο τη ε, έκθεση που έχω μπροστά μου είναι για τι 7 ε, Νοεμβρίου, ε, που σημαίνει. Μάλλον 17, με συγχωρείτε που ε, σημαίνει ότι μέχρι τις 15 πρέπει να έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες για να ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 24 Ιανουαρίου και να παρουσιαστεί το θέμα στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Ε, βεβαίως μπορεί να αναθεωρηθεί το χρονοδιάγραμμα, αλλά αυτή τη στιγμή έχει όπως όσα ανέφερα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, ε, στο υπαριθμό 7, είναι η έκθεση του κυρίου Κάζα για το μέλλον του ΦΠΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι περισσότερες τροπολογίες ήταν πολύ οικοδομητικές και χαίρομαι που βλέπω ότι ήδη υπάρχει συνένεση στα βασικά στοιχεία του μέλλοντος του ΦΠΑ. Κάποιες διαφορές ιδεολογίες όμως έχουν εμφανιστεί και αυτές αφορούσαν το βασικό ακόμα ρόλο του ΦΠΑ. Αφενός ε, βλέπουμε ε, το ΦΠΑ ως ε, εργαλείο πολιτικής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις κυβερνήσεις για να ανταποκριθεί σε άλλους στόχους, στόχους πολι... Ε, κοινωνικούς. Και άλλη άποψη είναι ότι θα πρέπει να επιβληθεί με ομοιομορφία έτσι ώστε να υπάρχει η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στο μεγαλύτερο βαθμό δυνατόν. Παρά τις διαφορές, οι διαπραγματεύσεις επί των ε, ε, συμφωνιών έχουν ξεκινήσει, έχουν τροχιοδρομηθεί και ελπίζω ότι θα βρούμε μια χρυσή τομή. Ε, τώρα, όταν αναφερόμαστε στις αιτολογικές σχέσεις, τα εισαγωγικά σημεία αναφέρονται σε διαφορά από την άμεση στην έμεση φορολογία. Αυτό δεν ήταν θέμα προτίμησης για τη μία ή την άλλη μορφή φορολόγησης, αλλά για να αναγνωρίσουμε μια τάση που υποδεικνύει στον μελλοντικό ρόλο του ΦΠΑ. Ε, καλωσορίζω τις τροπολογίες που έχουν αποσαφηνίσει αυτό το θέμα και υποστηρίζω τις τροπολογίες 1 έως 8, καθώς και 11 έως 13 και 15. Στην τροπολογία 9 τώρα, θα θεωρούσα ότι τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και τον ενεργειακό φόρο να είναι έμεσες και όχι άμεσες φορολογίες και ε, δέχομαι να ε, περιλάβω τις απόψεις που ε, είναι σε μια μορφή συμβαστικού κοινέμου. Δεν πρέπει να αναφερθεί ο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Είναι επίμαχο θέμα που δεν σχετίζεται με το ΦΠΑ και μπορεί να επισκιάσει τα πιο σημαντικά θέματα και θέλω να αποφύγουμε μια συζήτηση για το κατά πόσο θα υποστηρίζουμε ή όχι αυτό τον φόρο των χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών. Γι' αυτό αντιτίθεμαι στις τροπολογίες 14, 17 και 27. Τώρα, στον σχεδιασμό του ΦΠΑ καθορίζω την τροπολογία 16, 18 και 19 σχετικά με τη, τους μειωμένους σύντελεστές και τις απαλλαγές έχω παραδείγματα κάποιων ασυνεπιών και υπάρχουν αρκετές και θα υποστηρίζω την ουσία των τροπολογιών 20, 21, 24, 26 και 28 ε, με συμβιβαστικό κείμενο το οποίο θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα θέματα έχει ήδη κυκλοφορήσει ανάμεσα στους σκιώδεις εισηγητές. Μπορώ να δεχτώ τις τροπολογίες 22 και 23 με κάποιες ελαφρές αλλοιώσεις και την τοπολογία 25 και για την κατάργηση όλων των απαλλαγών και ε, του ε, μειωμένων συντελεστών, παρόλο που καταλαβαίνω την, το πνεύμα της τροπολογίας, η κατάργηση όλων των απαλλαγών ε, είναι κάπως υπερβολική. Γι' αυτό δεν θα υποστηρίξω αυτή την τροπολογία. Οι περισσότερες τροπολογίες υποδεικνύουν προς συνένεση για την πρόθεση αυτή της έκθεσης να αναγνωρίσει το status quo και ε, να πάμε στην αρχή του, ε, του, του ε, προορισμού. Φαίνεται να υπάρχει και συνένεση για το ότι αναγνωρίζεται η τάση προς σύγκληση εθνικών συντελεστών ΦΠΑ. Ένα συμβιβασμό είναι υποδιαπραγμάτευση για την αποσαφήνιση αυτών των παραγράφων. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που θέλουν να διαγράψουν αναφορά σε συγκεκριμένα ποσοστά και ε, θα αποδεχτώ την αφαίρεση αυτού του αριθμού. Και τέλος, ό,τι αφορά στον μείωση ε, της γραφειοκρατίας. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο έτσι ώστε να μην ε, γίνει το σύστημα ευπαθές στην απάτη. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Γι' αυτό έχουν ήδη κυκλοφορήσει συμβιβασμοί ε, σε αυτό το θέμα και καλωσορίζει την τροπολογία ε, που προσθέτει αξία στη συνήθισή μας μείωση της γραφειοκρατίας. Ιδιαίτερα καλωσορίζω τι τροπολογίες 49 και τροπολογία 54. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ίσως μπορούμε να είμαστε σύντομοι ε, και να κερδίσουμε λιγάκι χρόνο. Απευθύνομαι κυρίως στους και εισηγητές. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που επιτέλεσε και τις προσπάθειες που κατέβαλε για να συντάξει συμβιβαστικές τροπολογίες και προτάσεις που απηχούν τις απόψεις όλων μας. Πρόκειται για κάτι το σημαντικό για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η απλοποίηση κάποιων διοικητικών μεθόδων και μηχανισμών είναι πολύ αποτελεσματική. Είναι εξαιρετικές οι προτάσεις και υπάρχουν, πρέπει να πω, κάποιες προσαρμογές οι οποίες πρέπει να γίνουν για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. διότι βλέπουμε ότι εδώ συμπεριλαμβάνονται και θέματα πολύ σημαντικά, όπως ε, επιβολή ΦΠΑ στην ενέργεια ή στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί το θέμα του ΦΠΑ στα ενεργειακά προϊόντα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση και με την έκθεση που, της κυρία Λούλιν που εξετάσαμε και προηγουμένως. Θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί στον τρόπο προσέγγισης αυτού του θέματος. Τα διάφορα μέσα μεταφοράς επίσης είναι ένα, άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Τα, μιλώ για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα πρέπει να έχουν ένα ενιαίο ΦΠΑ και αναφέρομαι και στις εναέριες μεταφορές. Και να μην ξεχνούμε και την περιβαλλοντική πτυχή των μέσων μεταφοράς που πρέπει να προσέξουμε επίσης στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την πλήρη υλοποίηση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Το ότι θέλουμε παντού να κάνουμε πιο πράσινες πολιτικές, όπως λέγεται, είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πιστεύω επίσης ότι η συμβιβαστική πρόταση ΔΕΛΤΑ που αφορά το ίδιο θέμα είναι σημαντικό. Θα πρέπει κάποιες μειώσεις, κάποιες απαλλαγές να λάβουν υπόψη και τον κοινωνική πτυχή και την περιβαλλοντική πτυχή, αλλά να μην είμαστε πάντα πάρα πολύ περιοριστικοί σε αυτά τα οποία λέγουμε. Τέλος πάντων, για αυτές τις μικροδιαφορές που έχουμε, θα υποβάλουμε κάποιες συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Πιστεύω όμως ότι σε πολλά σημεία μπορούμε να συμφωνήσουμε και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, <clears throat> θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Νομίζω ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και τελικά θα πετύχουμε ευρεία συνέναση. Όπως ακούσαμε, εδώ πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Πιστεύω όμως ότι η προσέγγιση του εισηγητού είναι η σωστή κατεύθυνση ακόμα και αν ε, γνωρίζουμε ότι τελικά σε όλες τις χώρες υπάρχουν κάποιες αιρέσεις. Ο βασικός στόχος ε, πρέπει να είναι η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. Όμως ε, αν ε, οι εξαιρέσει ε, δεν εμποδίζουν την ε, δημιουργία της κοινή αγοράς, πρέπει να τις αποδεχτούμε. Στην αρχή, όταν ξεκίνησα στην πολιτική, ήμουνα απόλυτος και κάθετος όσον, αφορά, όσον αφορούσε τότε στο ΦΠΑ ε, τώρα όμως ε, που δεν ξέρω, έχω μεγαλώσει με πιο όριμος, ε, κατέληξα στο ότι αυτή η απόλυτη και κάθετη γραμμή δεν είναι ρεαλιστική. Ο κύριος Μπόλκενστάιν, ε, θυμόμαστε τι προσπάθησε να επιτύχει μερικά χρόνια και τελικά χτύπησε με το κεφάλι στον τοίχο. Το σύστημα λοιπόν είναι κατακαιρματισμένο και σε ορισμένες περιπτώσεις πράγματι δημιουργεί προσκόμματα στην κοινή αγορά. Γι' αυτό λοιπόν τον και θα πρέπει να κάνουμε. Εγώ υποστηρίζω και την ιδέα της ε, φορολογικής ε, ουδετερότητας. Οι εταιρείε δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο. Ε, ακούσαμε ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερος φορολογικός συντονισμός, αλλά ίσως όχι και απόλυτος. Εξακολουθεί να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει περιθώριο για φορολογικό ανταγωνισμό. Όχι να δημιουργούνται προβλήματα στα φορολογικά συστήματα, αλλά φαντάζομαι δεν θα εκπλαγείτε ή δεν εκπλήσεστε που εγώ ως φιλελεύθερος ομιλώ και περί ανταγωνισμού. Ο κύριος Βολφ Κλίντς, ε, ο συνάδελφός μου ε, που κάθε δεξιά μου, ε, έπρεπε να φύγει μια συνάντηση στη Γερμανία. Ήθελε όμως να υπογραμμίσει ότι το ΦΠΑ είναι μια πολύ σημαντική ε, φορολογική βάση, ε, τουλάχιστον ε, στη σημερινή εποχή. Ένα άλλο λοιπόν επιχείρημα για λιγότερες εξαιρέσεις είναι ότι οι Υπουργοί Οικονομικών χρειάζονται μια βιώσιμη και ακλόνητη βάση και το ΦΠΑ είναι ένα τέτοιο στοιχείο αποτελεί μία ακλόνητη βάση. Στη Γερμανία οι εξαιρέσει ε, ανέρχονται σε 20 δις ευρώ. Ελπίζω να είναι σωστό αυτό το στοιχείο που μας ε, ο συνάδελφός μου, αλλά αν ευσταθεί πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό. Ε, μπορούμε λοιπόν να έχουμε λιγότερες εξαιρέσεις και αυτό θα ήταν χρήσιμο. Τουλάχιστον οι Υπουργοί Οικονομικών θα ήταν ευτυχέστεροι. Πάω τώρα Στη δική μου την ερώτηση και ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ πρόκειται για την τροπολογία 40 και την υπαριθμό 56 και αυτές ε, οι τροπολογίες ε, υπογράφονται από μια σειρά συναδέλφων. Ε, δεν άκουσα, μάλιστα, εντάξει, τις στηρίζει αυτές τις τροπολογίες, αλλά δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν αρκετές χώρες που έχουν μειώσει το συντελεστή ΦΠΑ για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Και αυτό σχετίζεται και με αυτά που θα ζητήσουμε στην έκθεση του κυρίου Μπάλτς για τον αθλητισμό και σχετίζεται και με αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως για τα ε, στοιχήματα σε απευθεία σύνδεση. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με την χρηματοδότηση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών όπως είναι η ε, λέσχες ε, ποδοσφαίρου ή αεραστεχνικές μάλλον ε, που στηρίζουν τους ε, νέους παίκτες. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε από την Επιτροπή να είναι, λιγάκι, να είναι περισσότερο φιλελεύθερη. Δεν ξέρω κατά πόσον ο εκπρόσωπος της Κομισιόν το καταφέρνει, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί. Και αν εμείς στηρίξουμε αυτήν την ιδέα και ελπίζω ότι ο κύριος Κάζο, ο εισηγητής μας, ε, θα στηρίξει την ιδέα, ε, τότε φαντάζομαι ότι και η Επιτροπή θα ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τώρα το φόρο χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών, δεν ξέρω πόσες ώρες έχουμε συζητήσει για το φόρο αυτό. Πρέπει να ομολογήσω ότι εγώ δεν πίστευα ότι θα εφαρμοστεί ποτέ. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτές τις ε, τελευταίες ημέρε γίνονται τόσα πολλά πράγματα στην Ευρώπη που ίσω και αυτός ε, τελικά να... Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν νομίζω όμως ότι πρέπει η συζήτηση αυτή να γίνει σε αυτήν την έκθεση ε, να συμφωνήσουμε ότι η συζήτηση δεν ενδείκνυται σε αυτό το σημείο. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κάζα. Εγώ δεν στηρίζω αυτό το φόρο, πιστεύω ότι θα δημιουργήσει εμπόδια στην Ευρώπη, αλλά ίσως τελικά να επιβληθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας παρακαλώ πολύ, το θέμα αυτό του φόρου χρηματοψηφιακών συναλλαγών να παραμείνει εκτός αυτής της έκθεσης του κυρίου Κάζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Θα ευχαριστούσα τον κύριο Κάσα και το γραφείο του που συνέταξαν αυτή την σύντομη περιευτική έκθεση. Τα συστήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη διαφέρουν μεταξύ του και σε αποδοτικότητα και θα πρέπει να έχουμε ένα ευρύ πλαίσιο για ένα νέο σύστημα ΦΠΑ που να μειώνει τα λειτουργικά κόστη και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τις αρχές φορολογικές. Ένα αποδοτικό σύστημα που θα αυξήσει τα έσοδα, θα ενισχύσει την ενιαία αγορά και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Πρέπει να πω ότι έχω απογοητευτεί γιατί κάποιοι έχουν υποβάλει τροπολογίε που είναι εκτό του πεδίου εφαρμογής αυτής της έκθεσης. Θα πρέπει να αναπτύξουμε μία στρατηγική για το ΦΠΑ και ε, έχουμε απομακρυνθεί απομακρυνόμαστε από αυτό εάν κάνουμε μια, ένα κατάλογο επιθυμιών, και κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερο ανταγωνιστική από ό,τι είναι. Αν θέλουμε το Συμβούλιο να μας λάβει σοβαρά στα ε, υπόψη, θα πρέπει να έχουμε μια εστιασμένη ε, έκθεση στον ΦΠΑ. Χαίρομαι που ο κύριος Κάσα είπε ότι δεν θέλει η έκθεση να ασχοληθεί με τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και εγώ συμφωνώ με αυτό. ένα συνάδελφο είπε ότι υπάρχει ε, συνένεση για τον φόρο αυτό. Δεν πιστεύω να υπάρχει. Μπορεί στην Ευρωπτώνη να υπάρχει. Θα αν οι χώρε τη Ευρωζώνη ε, είχαν επιβάλει αυτό τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλογών διότι σημαίνει ότι θα μπορούσαν να κάνουν όλε τι επιχειρήσει του στο Λονδίνο αλλά αν δοκιμάσουμε να τον επιβάλλουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ε, βέβαια θα έχει το βέτο του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν έχει νόημα να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Χαίρομαι για τις αρχικούς ε, συμβιβασμούς που έχει υποβάλει ο κ. Κάσα και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί του. Ευχαριστώ. Ε, από τους φοράσινους ο Φιλίπ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομος. Συνήθως αρέσει να είναι εστιασμένες οι εκθέσεις και ε, συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι θα πρέπει να μην ξαναφέρουμε στην επιφάνεια τον φόρο χρηματοδοτικών συναλλαγών. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω και αυτό είναι ένα σύνδεσμο. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι κάποιες επιχειρήσεις ε, δεν καλύπτονται από τον ΦΠΑ δεν διαφεύγουν αλλά δεν καλύπτονται. Και ε, θα πρέπει να πούμε ότι σημειώνουμε ότι αυτή τη στιγμή οι χρηματοπιστωτικέ ε, υπηρεσίε δεν καλύπτονται από το ΦΠΑ και αυτό είναι ένα θέμα. Χωρί να πούμε πώ μπορούμε να το λύσουμε. Αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτέ οι, οι, οι υπηρεσίε δεν καλύπτονται. Και είναι ένα πρόβλημα γιατί είναι θέμα του ποια είναι η φορολογική βάση. Και γιατί επί ποιας βάσης μια τέτοια δραστηριότητα δεν πρέπει να υποβληθεί σε φορολογία σε σύγκριση με άλλες υπηρεσίες. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε γι' αυτό. Γι' αυτό ε, θα έπρεπε να κάνουμε μια αναφορά όπως κάνουμε και για τις αεροπορικές ε, ε, κοινωνίες. λοιπόν, γιατί, απαλλάσσεται, γιατί απαλλάσσονται σε αντίθεση με τις σιδηροδρομικές. Αυτό μπορεί να προκαλεί δια, στρέβλωση της αγοράς. Θέλω να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός. Βεβαίως. Αυτά ήταν τα σημεία που ήθελα να γύρω σε αυτές τις δύο απαλλαγές. Ε, βέβαια, αυτή δεν είναι έκθεση που αφορά τον φόρο επιχρηματοδοτικών συναλλαγών και δεν θέλω να επαναλάβω όλα τα επιχειρηματά που ακούστηκαν και θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε και στο εκείς μέλλον φυσικά, αλλά να υποδείξουμε ότι αυτή η δραστηριότητα ε, ξεφεύγει από την κάλυψη του ΦΠΑ και θα είναι καλά να το συμπεριλάβουμε. Ε, η διατύπωση μου για την διαγραφή των απαλλαγών και ίσως εκεί η διατύπωση να είναι κάπως φουνταμενταλιστική θα έλεγα, τα σημεία που ήθελα να γύρω είναι τα εξή. Συμφωνώ με τον Άσλι Φόξ. Όταν λες ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που είναι λιγότερο δαπανηρό για τους ε, φορολογούμενους αλλά και για τις φορολογικές αρχές. Συμφωνώ με αυτό. Και από αυτή την έννοια, αν απλουστεύσουμε το σύστημα και εδώ δι- το κάνουμε πιο εναρμονισμένο, αυτό βοηθάει. βοηθάει. Ε, αντιλαμβάνω αυτό που λες για την φορολογικό ανταγωνισμό. Όταν βλέπω όμως την κατάσταση όπου όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα φορολογικά έσοδα, ε, μπορεί ε, να συμφωνώ με το ποιος διαχειρίζεται καλύτερα το δημόσιο συμφέρον, αλλά για μένα αυτό που επήγει τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τα κατάλληλα και επαρκή φορολογικά έσοδα και γι' αυτό είναι καλύτερο να κάνουμε μια συνεργασία ή συντονισμό και όχι ανταγωνισμό. Και αυτό είναι θέμα επίγον και θα πρέπει να το τονίσουμε. Και έτσι ο συμβιβασμός που προτείνει ο David Κάζα αναφέρεται και στα δύο. Δηλαδή, θα πρέπει να συγκλίνουμε, αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν ταυτόχρονα και τη ε, δυνατότητα να διαφέρουν. Είναι, ε, δεν, δεν ξέρω ακριβώς ε, τι αναφέρεται εδώ, και μαύρο και άσπρο. Θα πρέπει ίσως να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι σε αυτό το θέμα για το τι επιθυμούμε. Αν τα καταφέρουμε να βρούμε μια συμφωνία, όπως λέω εγώ, η άποψή μας είναι ότι τους καιρούς μας αυτούς χρειαζόμαστε ένα ε, σύστημα που να συγκλίνει, βέβαια όχι 100% αλλά να πούμε ότι η προτεραιότητα είναι να υπάρχει σύγκληση. Σε ό,τι αφορά τώρα, συμφωνώ με αυτά που είπε ο Σαΐτ για το, για μειωμένο φόρο για περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Ε, δεν, αυτό που πρέπει να έχουμε θα πρέπει να δούμε αυτό τον φόρο κατανάλωσης έτσι ώστε να έχει κοινά αγαθά. Ε, για παράδειγμα, εάν οι κλιματικές αλλαγές είναι ένα κοινό αγαθό, η καταπολέμησή τους, τότε θα πρέπει να δούμε ε, απαλλαγές σε αυτό το θέμα. Το κλειδί είναι ότι θα πρέπει να μπορεί να αποδεικνύεται. Θα πρέπει να μπορούμε να, το, να καταμετρούμε το κοινό αγαθό που μπορεί να αποδοθεί με τη μείωση, ε, για παράδειγμα, σε περιβαλλοντικό τομέα. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε και αυτό θέλουμε να δούμε. Γι' αυτό είμαι έτοιμος να συζητήσουμε την διατύπωση του κειμένου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόρτας. Ε, Πάρα πολύ σύντομα, διότι εγώ δεν ήμουν σκιάδος τις έκθεσης αυτής. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση και δύο ερωτήσεις στον εισηγητή. Η παρατήρηση είναι η εξής. Μου φαίνεται ότι ο φόρος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν θα πρέπει να τεθεί στα πλαίσια της έκθεσης αυτής. Μου φαίνεται όμως ότι είναι σημαντική η αναφορά, κυρίως στην αναφορά στην τροπολογία 10 της τάσης που υπάρχει οι ε, άμεσοι φόροι να αντικατασταθούν από τους έμεσους. Και αυτό έχει μεγάλη σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα εδώ. Μετά από αυτά τα οποία ελέγχθησαν για τις τροπολογίες, νομίζω ότι μπορεί να βελτιωθεί η έκθεση και θα ήθελα να κάνω σε σχέση με το θέμα αυτό δύο ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν και αντικείμενο προφορικών τροπολογιών πριν να φτάσουμε στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Πρώτη ερώτηση είναι η εξή. Είναι κάτι το οποίο εμείς στα πορτογαλικά λέμε ΦΠΑ ταμείου. Τι εννοώ. Υπάρχει μία πρώτη τροπολογία που αναφέρεται, με την οποία δεν συμφωνώ, για απαλλαγή των ΜΜΕ. Νομίζω ότι είναι αποφασιστική σημασία για τις επιχειρήσεις να μην καταβάλουν ΦΠΑ στο κράτος πριν να το έχουν εισπράξει. Διότι διαφορετικά έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό συμβαίνει συνήθως. Πρέπει να πληρώνουν εκ των προτέρων το ΦΠΑ, να καταβάλουν εκ των προτέρων το ΦΠΑ στο κράτος. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη και σε αποτελέσει αντικείμενο προφορικής τροπολογίας. Και τελευταία ερώτηση παρατήρηση. Εγώ είμαι υπέρ του να Υπάρχει στρατηγική για την ριζική μείωση των ε, φορολογικών απαλλαγών ή μειώσεων, αλλά δεν υπάρχει καμία αναφορά στη δυνατότητα να υπάρξει βαρύτερη φορολογία σε κάποια άλλου είδους έσοδα. Νομίζω ότι θα πρέπει στα αγαθά πολυτελείας να επιβληθεί διαφορετικού είδους φορολογία. Διότι εμείς φορολογούμε με το ίδιο ΦΠΑ όλα τα προϊόντα και τα προϊόντα ε, ε, πολυτελείας δεν πρέπει να αποτελέσουν ειδικό αντικείμενο φορολόγησης. Θέλει κανένας άλλος συνάδελφος το λόγο. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί και εγώ πιστεύω ότι τελικά ε, μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία όσον αφορά την τελική ψηφοφορία. Ε, Θέλω όμως να πω ότι διαφωνώ με τον κύριο Πόρτας όσον αφορά στο να υπάρχει ένα κατόφλι εξαίρεσης ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για το 90% του συνόλου της ευρωπαϊκής οικονομίας και διότι ε, διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν ε, διαφορετικά όρια άρα δηλαδή ε, θα έπρεπε ίσως ε, να υπάρχει ε, κάποιο, κάποιο όριο σχετικά με τον νότιο όριο για να μην υπάρχει και ο, ο, ο ανταγωνισμός, ο αντισόπιτος ανταγωνισμός. Θα είμαι πολύ σύντομη κι εγώ γιατί νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην επόμενη έκθεση του κυρίου Μπάλτσα θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε λίγα πράγματα, να στηρίξω τους αδέλφους Λούτβιχ και Σμιτ ε, σχετικά με τις τροπολογίες που κατέθεσαν. Εδώ ε, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της έκθεσης και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την πράσινη βίβλο της Κομισιόν και την ψηφιακή ατζέντα που αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει σύγκληση σε όλους τους τομείς αλλά ε, κυρίως όσον αφορά τα ηλεκτρονικά βιβλίο ε, και τις ε, εφημερίδες. Ίσως ο εισηγητής μπορεί να αφαιρθεί ιδιαίτερα στο θέμα αυτό. Και πολύ σύντομα να πω σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε για το ευρύτερο πλαίσιο. Συμφωνώ και εκτιμώ τη δουλειά του εισηγητή που προσπαθεί να βρει συμβαστική πρόταση κυρίως όσον αφορά στις τροπές σχετικά με τις ε, εξαιρέσει και την ευελιξία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Εξετάζουμε τις εξαιρέσει σε σχέση με την ευελιξία. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να υπάρχει ευελιξία ε, για λόγου δημόσια πολιτική. σε βαθμό βέβαια που ε, δικαιολογείται κάτι τέτοιο. Ίσως θα πρέπει σε αυτή τη σημαντική πρόταση να φέρονται κάποιε ρήτρε αιτιολόγηση. Υπάρχουν παραδείγματα κυρίως για περίοδο ε, οικονομικής ύφεσης. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, στην προηγούμενη κυβέρνηση καταβήκαμε στο 17,5 ΦΠΑ μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτή ήταν η ευελιξία μας και το κάναμε αυτό για να τονώσουμε την κατανάλωση. Οι συντηρητικοί ανέβασαν το συντελεστή στο 20% και αυτό είχε αντικές επιπτώσεις στην οικονομία και στον καταναλωτή. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι τρόποι εσόδων. Ε, κατόπιν τούτου δεν πρέπει να υπονομεύσουμε υπερβολικά την ευελιξία. Όπως σας είπα, ίσως θα πρέπει να δούμε τις εξαιρέσεις, αλλά να αναφέρουμε και τις αιτιολογίες, αιτιολογημένες εξαιρέσεις και όχι να ανοίξουμε διάπλατα την πόρτα σε ε, κάθε μορφή εξαίρεσης. Δεν ξέρω μήπως ε, η Κομισιόν ε, θέλει το λόγο. Όχι. Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους, ε, για τις προτάσεις τους. Οι περισσότερες προτάσεις έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις ε, τροπολογίες, στις συμβαστικές που διένυμα σήμερα το πρωί. Άρα δηλαδή οι συνάδελφοι θα έχουν αρκετό χρόνο για να εξετάσουν τις συμβαστικές προτάσεις. Και βεβαίως εξαιρείται το θέμα του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όλες οι άλλες απόψεις ε, πρέπει να πω ότι σε μεγάλο βαθμό συμπεριλήφθηκαν στις ε, αρχικές μου τροπολογίες. Και λίγα μονολόγια όσον αφορά την ε, τροπολογία υπερθών 14 έγινε αυτή αποδεκτή και ως προς την αποτελεσματικότητα ε, συλλογής ε, εσόδων από ΦΠΑ υπάρχει εδώ συνένεση και πρόκειται να συντάξουμε μια διαφορετική συμβαστική τροπολογία όπου θα αναφέρονται τα θέματα κατά προτεραιότητα. Όσον αφορά τώρα τη νομική διαδικασία, συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή τα νομικά εργαλεία περιλαμβάνουν και ασαφείς διατάξεις, αλλά δηλαδή και εκεί πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Και με μεγάλη μου χαρά στηρίζω την τροπολογία 68 που ε, προσθέτει αξία μέχρι την ε, ψηφοφορία που θα γίνει κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο. Έχουμε ακόμα χρόνο στη διάθεσή μας. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τους ε, συναντέλφους μου για να βρούμε κάποια ισορροπία όπου αυτό ε, κριθεί απαραίτητο. Πράγματι θα ψηφίσουμε στις 19 Σεπτεμβρίου για να πάει το θέμα στη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Και πάμε τώρα στην επόμενη έκθεση στην έκθεση του κυρίου Μπουκχάτ ε, Μπάλτς. Αν χρειαστεί θα συζητήσουμε το θέμα αυτό μέχρι τις 12.30 και το επόμενο θέμα του κυρίου Μπάλτς θα πάει για ε, σήμερα το απόγευμα μετά τις ψηφοφορίες όπου θα έχουμε χρόνο. Μπουκχάτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στο σχέδιο της έκθεσης για την οδηγία αυτή ε, έχω κατ' ουσίαν εφαρμόσει αυτά τα οποία είπαμε στις 21 Μαρτίου. Πάρα πολλές ε, τροπολογίες είναι τεχνικής φύσεως, ε, οι οποίες απορρέουν από την οδηγία Solvency 2 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της στις αρχές αυτού του έτους ε, έθεσε σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τον κανονισμό για τις ασφάλειες. Για μένα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η προσαρμογή των επιτοκίων ε, κυρίως όταν πρόκειται για προβλήματα ρευστότητας ε, στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ένα άλλο θέμα που έχει σημασία είναι η ισοτιμία τρίτων χωρών και ε, μια μεταβατική διάταξη, κάτι το οποίο έχει εφαρμόσει ευρέως η Κομισιόν για να αποφύγει κατά την άποψή μου τη συγκεκριμενοποίηση. Βεβαίως οι συζητήσεις ε, δεν απλουστεύονται με την ε, Omnibus του οδηγία αλλά και με τα εφαρμοστικά μέτρα. Έτσι λοιπόν είχαμε την σχετική μελέτη όταν κατατέθηκε η σχετική οδηγία για την οδηγία Omnibus 2. Ε, αυτό δεν το αναφέρω τόσο ως κριτική, όσο περισσότερο ως διαπίστωση. Τέλος, θεωρώ ότι στο Συμβούλιο ε, βλέπουμε ότι ο καθένα ε, προσπαθεί να προβάλλει τα δικά του συμφέροντα. Όλοι διεκδικούν ένα κομμάτι από την πίτα, άλλοι μεγαλύτερο, άλλη μικρότερο και μόλις κάποιος ε, έχει στο χέρι του το πιάτο που θα βάλει το κομμάτι της πίτας, τότε μοιάζει να πλησιάζουμε και στην τελική λύση. Εγώ ε, παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις ε, στο Συμβούλιο, αλλά πρέπει να σας πω ότι καταρχήν ε, πρέπει να πιστώ για το ότι πρέπει να βρούμε κάποια λύση που θα είναι αποτελεσματική για την αγορά. Αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο ε, προσπαθεί να βρει κάποιες αλλαγές, matching premium, ε, αντικυκλικό ε, για αυτά τα δύο τουλάχιστον είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Στις δικές μου τις προτάσεις περιλαμβάνω την ενίσχυση ε, της εποπτείας ε, επί των ασφαλιών στην Ευρώπη. Κυρίως κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπου δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές περιεχομένου, ε, οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο της οδηγίας πλαίσιο. Γιατί και οι εποπτικές αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν το στομότερο δυνατόν ασφάλεια για τις νομικές ρυθμίσεις που θα επέλθουν. Όσον αφορά στα εφαρμοστικά μέτρα δεν μπορούμε να έχουμε μόνο πράξεις κατ' εξουσιοδότηση κυρίως όταν πρόκειται για θέματα ε, τα οποία χρίζουν της ε, τεχνογνωσίας ε, των εποπτικών αρχών. Είχαμε ε, την πρώτη οδηγία, Omnibus One, την οποία έχουμε ήδη εγκρίνει και σύμφωνα με αυτήν θα πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις ε, οι οποίες ε, θα επιφέρουν ασφάλεια στην αγορά. Όσον αφορά στις προδιαγραφές αυτές, θα πρέπει να ξανασυμφωνήσω με τον φορέα ΕΙΟΠΑ. Αυτό που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, μιλάω πάρα πολύ γρήγορα οι διερμηνείς ε, διαμαρτυρήθηκαν αγωνίζονται, λέει η πρόεδρο, να σα παρακολουθήσουν. Ο μιλητής και εγώ θέλησα να μιλήσω λίγο πιο γρήγορα για να υπάρχει χρόνος. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μιλήσω σε κάποιο πιο βραδύ ρυθμό. Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ε, ρύθμισης περιρευστότητας ε, τις ε, οδηγίες αυτέ να τι λάβουμε σοβαρά υπόψη μα. Και ε, επίση και τον φορέα ΟΙΟΠΑ. Σε τελική ανάλυση πρόκειται εδώ για ένα εργαλείο ε, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τεχνικών αποθεμάτων. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος που θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του πριμ. Και το πριμ θα πρέπει να καταβάλλεται μόνο σε περίπτωση έλλειψης ρευστότητας, κυρίως ε, για να αντιμετωπίσει κανείς ε, τα λάθη υπολογισμού που έχουν λάβει χώρα και επίσης ε, όταν οι αρμόδιες αρχές του κράτους εγκρίνουν αυτό το πριμ στους ασφαλιστές και στους αντασφαλιστές. Όσον αφορά τώρα τις ε, τρίτες χώρες, εγώ ε, τάσομαι υπέρ της ε, προσωρινής ισοτιμίας, δηλαδή τα τρίτα κράτη δεν θα παίρνουν απεριόριστες παραχωρήσεις όπως είχε αρχικά προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για αυτή την προσωρινή ισοτιμία, για να υπάρξει αυτή θα πρέπει να κατατεθεί και ένας ε, σχετικός κατάλογος. Νομίζω με τον τρόπο αυτό, ε, στη τελική ανάλυση, δίνουμε ισότιμα δικαιώματα στα τρίτα κράτη, ε, τουλάχιστον για πέντε χρόνια. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνονται πολλές μεταβατικές διατάξεις, όπου βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μεταθέσει πάρα πολλές νομικές πράξεις σε κατεξουσιοδότηση πράξης οι προθεσμίες αναφέρονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ τάσομαι υπέρ μιας, ενός μεταβατικού σχεδίου δύο σταδίων το οποίο θα πρέπει να παγιωθεί με την οδηγία πλαίσιο. Η οδηγία Solvency 2 όπως προβλέπετε θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε εθνικό δίκαιο από τον Ιανουάριο και εντεύθεν. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει προετοιμασία όχι μόνο των ασφαλιστικών εταιριών αλλά και των εποπτικών αρχών. Οι πληροφορίες για την εφαρμογή της Solvency 2 θα πρέπει να δουτούν ήδη στις εποπτικές αρχές γιατί ε, μέχρι τότε θα ισχύουν οι διατάξεις του Solvency 1. Ε, εγώ θεωρώ ότι κυρίως όσον αφορά τη διάρκεια του ενός έτους ε, η σχέση κόστους κόστους-οφέλους δεν είναι σωστή. Η επεξεργασία πληροφοριών ε, για μένα είναι πολύ σημαντική. Βεβαίως συμφωνώ απόλυτα με το Συμβούλιο ότι το έτος 2013 πρέπει να το εκμεταλλευτούμε για αντιοδοτήσεις, ε, κυρίως όσον αφορά το περίφημο εσωτερικό μοντέλο. Την 1η Ιανουαρίου του 2014 η εφαρμογή του Solvency 2 ε, θα υπάρχει πλέον με συνοδευτικά μέτρα. Και έτσι λοιπόν για δύο, κράτη, ένα, για δύο χρόνια ένα κράτος ε, θα μπορεί ε, σε ασφαλιστικές εταιρείε, μικρές και μεγάλες, στην περίπτωση που δεν καλύπτουν το κεφάλαιο προβλέπεται στη Solvency 2, να τους χορηγεί μία ε, μεταβατική περίοδο το ε, όριο για, τα όρια για τα ελάχιστα κεφάλαια θα πρέπει προφανώς και να τηρούνται και θα πρέπει να κατατίθενται και οι σχετικές εκτέσεις περί πρόοδου. Εγώ είμαι υπέρ μιας ε, μεταβατικής περίοδου 10 ετών για υβριδιακά κεφάλαια και για τα repackage loans. Συμφωνώ με αυτό. Να υπάρχει ε, μια συνεργασία με τις τράπεζες. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο κατά την άποψή μου είναι ένα software που να ε, μπορεί να χρησιμεύσει για τη μετάβαση και εδώ προτείνω ε, μεταβατική περίοδο διάρκειας δύο ετών ε, κατά την οποία περίοδο θα εκμεταλλευτούμε τα ήδη υπάρχοντα συστήματα. Και εδώ έχω κατά νου κυρίως τις μικρές και τις μεσαίες ασφαλιστικές εταιρείες. Οι εφαρμοστικές διατάξεις θα υπάρξουν το 2012, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει στις εταιρείε που έχουν κάποιο πρόβλημα να του χορηγήσουμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να προετοιμαστούν καλύτερα. Όσον αφορά τις ε, μικρές ε, και τις ε, μεσαίες ασφαλιστικές εταιρείες, είναι σημαντικό για μένα να ενισχυθεί η αναλογική αρχή. Πιστεύω λοιπόν ότι το σχέδιο της έκθεσης ε, έχει να προσφέρει πάρα πολλά, αλλά έχοντας κατά νου τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, θα ήθελα να περιστώ σε αυτά τα σημαντικά για μένα θέματα. Κατόπιν τούτου σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω τις ε, πρώτες εκτιμήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι ο Έτβερτ θα μιλήσει εκ μέρους του Πίτερ Σκίνερ. Ο Πίτερ Σκίνερ, ο ασκιώδης εισηγητής, ε, ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να παραβρεθεί. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μπάλτς για αυτή την έκθεση, την προσχέδιο έκθεση της Omnibus 2 τώρα το, μπαίνουμε στην περίοδο τροπολογιών και πέραν από αυτή. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ντοσχέ τεχνικών ε, λεπτομεριών, αλλά είναι και ένα ε, κουτί εργαλείων, ρυθμιστικών εργαλείων και θα πρέπει να αποδείξουμε μια συνεχτική και περιεκτική ε, προσέγγιση γιατί η οδηγία Φρενγκιότητα 2 είναι πρωταρχικό μας μέλημα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προχωρήσουμε έτσι ώστε αυτό το τι εργαλείων ενισχύεται. Έχουμε τρία σημεία, τονίζουμε. Πρώτον, οι νομικές ε, εξουσίες που δίνονται στον ΕΙΟΠΑ και επίσης ε, το πρίμα Σχετικά με τα νομικά θέματα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν παραβιάζουμε ε, τον, την απόφαση Μερώνη και η ΟΠΑ δεν ε, ε, υπερτερεί τη δικής της νομοθεσίας. Θα πρέπει να δώσουμε στην αρχή η ΟΠΑ τα, εργαλεία που χρειάζεται. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε το θέμα της ισοτιμίας. Ε, καθώς επιβάλλεται η Solvency 2 θα πρέπει να συνεχίσουμε να βλέπουμε τα μέσα με τα οποία οι τρίτες χώρες μπορούν να ε, προσαρμοστούν στο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δομή μας θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε χώρες που έχουν συναλλαγές στα σύνορά μας και, ε, και των ασφαλιστών μας που κάνουν επιχειρήσεις εκτός. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με το περίμα ρευστότητα. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό εργαλείο για τους ασφαλιστές να χρησιμοποιούν ε, σε ε, περιπτώσει προβλημάτων στις αγορές. Αυτές οι δύο έννοιε θα πρέπει να υλοποιηθούν με τρόπο που να συνάδει με το νομικό προηγούμενο. Και πάλι συγχαίρω τον κύριο Μπάλτ και ε, θα συνεργαστούμε με όλους τους άλλους σκιώδεις σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο σκιώδης ε, των Άλτε είναι η Σεβίγκουλα που δεν βρίσκεται εδώ ε, και ήμουν και εγώ σκιώδης στη Solvency 2. Υπάρχουν τρία θέματα τα οποία θέλω να γύρω και βέβαια έχουν σχέση, στενή σχέση με τα τρία θέματα τα οποία έχουν αναφερθεί εκ μέρους του κυρίου Σκίνερ. Το πρώτο uh, uh, είναι το σημείο ε, των ατελών επιχειρήσεων και το πριμ ρευστότητας και τι, πώς σχετίζεται με τις μακροχρόνιες επενδύσεις. Και ήθελα πάντα να βρούμε μια λύση στο θέμα των ιδίων κεφαλαίων και αλλά γίνεται το θέμα του πώς θα το λύσουμε εάν και θα πρέπει να καθορίσουμε ότι θα βρούμε λύσεις σίγουρα σε αυτά τα ζητήματα και να το προδιαγράψουμε σε ένα στάδιο επίπεδου 1. Και μετά έχουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες και της αρχής ΕΙΟΠΑ και αυτό έχει αναφερθεί και την έγκριση των τοπικών ε, εποπτικών αρχών. Και εδώ ε, φτάνω στο δεύτερο θέμα που είναι αλληλένδετο των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων. Στην Solvency 2 αφήσαμε κάποιες ε, ατελείς υποθέσεις στις κατεξουσιοδότηση πράξεις ε, που δεν είχαμε το χρόνο να ανταποκριθούμε, δύο μήνες συν δύο μήνες είχαμε και ε, συνειδητοποιήσαμε ότι θα είχαμε ένα κείμενο 500 σελίδων το οποίο πρέπει να εξετάσουμε και και γι' αυτό είπαμε ε, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν μπορούμε να μην έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας. Ε, γι' αυτό ε, επίμεινα να έχουμε τρεις μήνες και τρεις μήνες και έχω συνεχείς αγώνες με την Επιτροπή στο θέμα αυτό και νομίζω αυτό είναι σωστό. Καθώς προχωρούμε, κάτι άλλο που συμβαίνει είναι ότι Έχουμε πάμπολες πράξεις κάτι εξουσιοδότηση που καταφάνουν και ε, συνειδητοποιούμε ότι χρειαζόμαστε το χρόνο στη διάθεσή μας και αυτό είναι σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε τι κάναμε όταν είχαμε εφεύρει του ρυθμιστικού τεχνικού κανόνε στην Omnibus 1, στη Γενική Οδηγία 1. Το σκεπτικό που είχαμε στο Κοινοβούλιο αρχικά ήταν ότι θέλαμε ε, να είναι πολύ ε, δυνατά αυτά και να μπορούμε να κάνουμε τεχνικά θέματα χωρίς οποιαδήποτε πολιτική παρεμβολή, διότι θα έκαναν πράγματα τεχνικά και οι αρχικές μας σκέψεις θα ήταν να ε, ξεπεράσουμε την Επιτροπή και Ανακαλύψαμε όμως ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει νομικός, γι' αυτό εφήβραμε τους λεγόμενους ρυθμιστικούς τεχνικούς κανόνες ως μια διαδικασία εξυγχρονισμού και τότε κάναμε ε, σε διάρκεια ενός μηνός συν ένα μήνα. Πρέπει να πω ότι τώρα ανησυχώ λίγο για το αν θα βρεθούμε ε, μπροστά από αυτό στις 500 σελίδες και σκέφτηκα ε, δύο μήνες συν δύο μήνες δεν ήταν αρκετή και ήθελα τρεις συν τρία και ε, δεν θέλω όμως να βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα έχουμε μόνο ένα μήνα συν ένα. Αναγνωρίζω ότι κάποια από τα πράγματα όμως επί συνεχή βάση που που θα συνεχίσουν θα ρυθμιστούν μέσα από τους ρυθμιστικούς τεχνικούς κανόνες και αυτό το, το ακόμη στη σκέψη μου και ε, δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε ότι την πρώτη φορά όταν έχουμε τις 500 σελίδες θα πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο διότι έχουμε πολλά πράγματα να επεξεργαστούμε ταυτόχρονα και ίσως στην αρχή, στην εκκίνηση θα πρέπει να είναι κατεξουσιοδότηση πράξη αλλά μετά ε, να περάσουν σε ρυθμιστικούς τεχνικούς κανόνες. Αρχίζω να το επεξεργάζομαι στη σκέψη με αυτό και σκέφτηκα ότι αξίζει να το αναφέρουμε και να πούμε και ποιο ήταν το σκεπτικό. Γιατί είχαμε την βραχύτερη περίοδο για... και βέβαια μαζί με αυτή την βραχύτερη περίοδο για τους ρυθμιστικούς τεχνικούς κανόνες ε, η ρυθμιστική αρχή, η ΕΙΟΠΑ, περιορίζεται, όπως αναφέρθηκε από τον Έντουαρτ, ε, στα πλαίσια της απόφασης Μωρώνη ότι δεν πρέπει να, ε, είναι, να έχει πολιτική χρειά. Και θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία εδώ, να δούμε ακριβώς ότι θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Θα πρέπει να γίνει περαιτέρω συζήτηση εντός της Επιτροπής, ε, γιατί το τελευταίο που θέλουμε είναι να μην έχουμε επιλογή ε, μπροστά μας και να καταλήξουμε σε ένα ρυθμιστικό τεχνικό κανόνα γιατί δεν είχαμε το χρόνο απλά και μόνο. Θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό που θα το στείλουμε πίσω και θα το ξαναδούμε για άλλους δύο μήνες. Διότι ε, βέβαια δεν είναι και πολύ σωστός τρόπος να χειριζόμαστε ε, τα πράγματα. Το, τρίτο, το τελευταίο σημείο είναι το θέμα της τρίτης χώρας. Είναι πολύ σημαντικό, εκ μέρους ε, του Πίτερ, ο Έντουαρτ ανέφερε ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτές οι τρίτες χώρες και οι συμφωνίες τρίτων χωρών λειτουργούν και εντός και εκτός. Εστιαζόμαστε σε αυτό που θέλουμε εμείς στην Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε δημιουργήσει ένα πεδίο ε, ε, δυναμικό όπου πρέπει όλοι να Υποάλλουν τους κανόνες μας εδώ στην Ευρώπη. Θα πρέπει όμως οι εταιρείε μας να είναι ασφαλείς γιατί ε, ακολουθούν τους κανόνες μας και εκεί που βρίσκονται. Αλλά τι γίνεται με τις άλλες εταιρείες που βρίσκονται εκτός της ομάδας που μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστικές γιατί παίζουν με βάση διαφορετικούς κανόνες. Ίσως αυτό προσπαθεί ο εισηγητής να εξετάσει με την ε, με προσωρινή αναγνώριση. Δεν είμαι βέβαια πώς θα εξελιχθεί μέσα στα πέντε χρόνια, διότι οι αγορές ε, εξτάζουν τα πράγματα σε πενταετής περιόδους. Προσπαθήσατε όμως να είστε καινοτόμο σε αυτό που προτείνετε και ίσως να είναι το καλύτερο που μπορούμε να προσφέρουμε αυτή τη στιγμή, διότι είναι ένα καθόδες πρόβλημα αυτό, είναι δύσκολο. Σας ευχαριστώ για το έργο σας και νομίζω θα είναι χρήσιμο για μας να συνεχίσουμε τη συζήτηση για να δούμε αν υπάρχει τρόπος να βελτιώσουμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση ή αν πρέπει να περιμένουμε να έχουμε αυτό το ενδιάμεσο μέτρο και να ε, αναφέρουμε ότι ε, στο τέλος αυτής της πενταετούς περίοδου ε, δεν θα καταλήξουμε σε μεγάλες δυσκολίες. Θα, είμαι βέβαια ότι θα δω και άλλα σημεία στην πορεία, ίσως και άλλα μέλη της ομάδας, γιατί εδώ Μιλάω και ως προεδρεύουσα και ως ε, σκιώδης και όχι εκ μέρους της ομάδας. Το επόμενο άτομο στον κατάλογο είναι ο κ. Έπινγκ από την ECR, ο Άσλι. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάλτ για αυτή την έκθεση. Σε αυτό το πολύ τεχνική φύσεω θέμα είναι σημαντικό να θεσπίσουμε τι κατεξουσιοδότηση υπεράξει και τα τεχνικά, του τεχνικού κανόνε, το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε οι ασφαλιστέ να είναι έτοιμοι για την ημερομηνία υλοποίηση. Και χαίρομαι που ο κύριο Μπάλτ αναγνώρισε ότι οι ημερομηνίε είναι κάπω φιλόδοξε και έκανε τροπολογίε για την σταδιακή υλοποίηση. Το υποστηρίζουμε, αλλά πρέπει να συζητήσουμε και τι λεπτομέρειε. Χαίρομαι που ο κύριο έχει κάποιες τροπολογίες σχετικά με την αναφορά, ιδιαίτερα τι σπεριτες απαιτήσει της αναφοράς γραμμή προς γραμμή των ε, περιουσιακών στοιχείων των ασφαλιστικών. Τώρα, ε, χαιρετίζουμε την προσωρινή ε, ισοδυναμία χρειαζόμαστε αυτές τις προσωρινές διευθετήσεις ε, από την περίοδο ανάμεσα στην ε, υλοποίηση στην Ευρώπη και την υλοποίηση σε άλλες δικαιοδοσίες. Αν δεν το κάνουμε αυτό θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις με τρίτες χώρες στην ουσία. Ήθελα να αναφέρω στον κύριο Μπάλτς τη δυνατότητα ότι αυτό το όριο των πέντε ετών μπορεί να μην είναι αρκετό και μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες θα πρέπει να παραταθεί αυτό το όριο. Επίσης υποστηρίζω τις τροπολογίες του κ. σχετικά με το συντελεστή έκπτωση και το πρίμα ρευστότητα. Θα πρέπει να γίνει μια διασαφήνιση της φόρμουλας και τον ορισμό του τι σημαίνει stressed market. Ωστόσο, η χρήση των κατεξουσιδότητων παράξεων ε, είναι ε, σημαντική για να έχουμε ε, τη σωστή πολιτική ενόραση θα πρέπει να αποφασιστεί πότε θα ε, χρησιμοποιηθεί ε, ο συντελεστής ε, έκπτωση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπάλτ και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί του. Ευχαριστώ για του πράσινου. Χαίρομαι πάρα πολύ που στο πλαίσιο του εξευρωπαϊσμού ε, των ρυθμίσεων για τις εποπτικές αρχές κάνουμε ήδη το πρώτο βήμα. Ο κύριος Μπάλτς αναγκάστηκε να περιμένει πάρα πολύ μέχρι να μπορέσει να ψάξει όλο αυτό το υποδόμημα που είναι πολύ περίπλοκο. Κατατέθηκαν πάρα πολλές τροπολογίες και νομίζω ότι χρειάστηκε και μεγάλος όγκος δουλειάς για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Πάντως η έκθεση αυτή ε, μπορεί να χρησιμεύσει για να εξάγει κανείς κάποια μαθήματα από την κρίση. Και ε, επιτρέψτε μου να φέρω κάποια σημεία. Το πρώτο είναι το εξής. Αφενός ε, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε πάρα πολύ για την επιρροή των οίκων αξιολόγησης στον χρηματοψηφιστικό τομέα και λέμε ότι πρέπει να αποδυναμωθεί ο ρόλος του. Το 9α εκεί η οδηγία Omnibus αναφέρεται στους οίκους αξιολόγησης. Ε, κατά την άποψή μας όμως όλο αυτό είναι αμφίσιμο. Πολύ και σωστό αυτό που λέει ο Μιλτής ότι πρέπει να υπάρχει ενίσχυση των υποπτικών, της εποπτικής αρχής ΑΙΟΠΑ. Όμως ε, ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τη δική μας την απόφαση. Δηλαδή τους οίκους αξιολόγησης και τις επιπτώσεις τους, κυρίως την επιρροή τους, να προσπαθήσουμε να την επιρροήσουμε, περιορίσουμε. με την οδηγία Solve έχουμε πλέον τα κριτήρια, αναφέρουμε στο άρθρο 75 της Συμφωνίας Solvency 2 και εκεί πρέπει να υπάρχει κάποια προσοχή, διότι αυτή η προκυκλικότητα μπορεί να ενισχυθεί. Ε, αυτό εμείς το επικρίνουμε κυρίως όσον αφορά θέματα λογιστικής στον τομέα των ασφαλιών ε, αλλά κυρίως ε, στον τομέα των ε, τραπεζών δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει η αξιολόγηση σε σχέση με την αγορά. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα που τίθεται είναι μήπως χρειαζόμαστε και άλλες μεθόδους αξιολόγησης για να αποδυναμώσουμε αυτή τη νέα ρύθμιση. Το τρίτο που θέλω να πω είναι, μιλάμε πάρα πολύ για κρατικά και δημόσια χρέη. Όμως στον τομέα των ασφαλιών εκεί δεν προβλέπεται η αντιμετώπιση των κινδύνων, sovereign Risks. Ε, σωστό είναι αυτό, τη στιγμή που υπάρχει κρίση. Ε, πάρα πολλοί γνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα με, τις, με την κεφαλαϊκή επάρκεια. Κατόπιν, ε, πολλοί θέτουν το θέμα των δύο κεφαλαίων στον τομέα των ασφαλιών. Έχουμε κεφάλαιο επίπεδου tier 3, στις ασφάλειες μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αυστηρά κριτήρια. Μόνο για τις τράπεζες. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να προτείνουμε κάτι τέτοιο ε, και στον τομέα των τραπεζών ε, tier 4 σε αυτό το επίπεδο μιλάμε για ε, νομισματικά κίνητρα για να υπάρχει ε, clearing στις τράπεζες όμως και οι ασφάλειες χρησιμοποιούν την αγορά των παραγόγων. Άρα δηλαδή δεν θα πρέπει και σε αυτόν τον τομέα να υπάρχουν σχετικές προβλέψεις για να υπάρχουν και κίνητρα για clearing χρησιμοποιούμε τις ε, προτάσεις του, μάλλον χαιρετίζουμε τις προτάσεις του εισηγητή σχετικά με την υποπτική αρχή ΑΙΟΠΑ. Επίσης ε, κάποιες από τις κατεξοδότητες πράξεις πρέπει να γίνουν τεχνικοί ρυθμιστικοί κανόνες. Σωστά όλα αυτά, όμως πρέπει να διερωτηθούμε μήπως με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση. Δηλαδή ένα τμήμα των στάνταρτ ε, θα έρθει ως κατεξοδότηση πράξη και ένα άλλο τμήμα θα έρθει ως ρυθμιστικός κανόνας. Με τον τρόπο αυτό όμως θα υπάρξει επιβράδυνση και ίσως ε, το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί με το να αποδίδουμε σημασία μόνο στις ε, τεχνικές ε, προδιαγραφές και να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Πάω τώρα στο πριμ έλλειψης ρευστότητας. Εδώ βλέπουμε ότι αυτό αφορά κυρίως τον ασφαλιστή και με τον τρόπο αυτό τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ασφαλιζεμένων. Ένας αντικυκλικός μηχανισμός στο Solvency 1, κάτι το οποίο έκανε το Συμβουλίο με το Prim Counter Cyclical, ε, μπορεί αυτό να γίνει, όμως ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να οδηγεί στο να αγνοείται η ε, κεφαλαϊκή ανεπάρκεια. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτό το Prim έλλειψης ρευστότητας. Οι ε, περιορισμοί που αναφέρει ο συγητής ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση, όμως νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Επιπλέον ε, πρέπει να αποφύγουμε σε επίπεδο 2 να υπάρξει ε, περαιτέρω άμβλυνση ε, των υφιστάμενων κανόνων. Όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις πρέπει να πούμε το εξής. Ε, το αρχικό σχέδιο θα συνεπάγεται μία σειρά ρητρών ανοίγματο. Ο εισηγητής πολύ σωστά λέει ότι όλα αυτά πρέπει να επανέλθουν στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και πράγματι ήταν απαραίτητο να υπάρξουν τροπολογίες και διορθώσεις για να μπορεί κανείς να διαβάσει καταρχήν αυτό το κείμενο. Και αυτό ε, που τέλο πάντων μπορούμε να το διαβάσουμε το οφείλουμε στον εισηγητή. Ε, κατά μέρο μας εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά θέματα. Πρώτον, το βρίσκουμε σωστό ε, κατά την εφαρμογή να προσφέρεται περισσότερος χρόνος. Εμείς προτείνουμε να υπάρχει και μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεγεθών. Μέχρι τώρα το όριο ήταν στα 5 δις αυτό όμως αφορά τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ίσως στις πολύ μικρές μπορεί κανείς να προσφέρει περισσότερο χρόνο και κατόπιν να εξετάσουμε το θέμα της κλιμάκωσης. Σε γενικές γραμμές εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιε μεταβατικέ διατάξει για τα ευρυδιακά κεφάλαια. Ξέρουμε ότι κάποιε ασφαλιστικέ εταιρείε ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα κεφάλαια αυτά, αλλά ανησυχούμε για το θέμα των μεγάλων μεταβατικών ρυθμίσεων. Και τι γίνεται τώρα, ορισμένε ασφαλιστικέ εταιρείε εκδίδουν ε, τέτοιο ή τέτοιου είδου κεφάλαιο, όχι μόνο για να προστατεύσουν αυτά που ήδη έχουν, αλλά κυρίω διότι πιστεύουν ότι μετά από 10 χρόνια ε, θα μπορέσουν να εκδώσουν ε, και άλλες, άλλους τέτοιους τίτλους να συγκεντρώσουν τέτοιου είδους κεφάλαια. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι βοηθάει τη ρύθμιση. Ε, κατόπιν άρθρο 111M. Εκεί προβλέπεται μια ειδική ρύθμιση, δηλαδή την αξιολόγηση των ε, συμμετοχών. Εκεί ε, στην αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να υπάρχουν χαμηλότερες απαιτήσει. Όμως αυτό ανοίγει τον δρόμο στο αρμπιτράζ. Και δεν ξέρω κατά πόσον αυτό εξυπηρετεί την πολύ καλή αρχή που εισαγάγατε ε, εσεί και που λέτε ότι είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στι ειδικέ ρυθμίσει. σω και εδώ ε, είναι μια τέτοια περίπτωση. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τι ε, τροπολογίε 26 και τι επόμενε. Αυτό αφορά στην οδηγία διαμεσολάβηση. Σωστά αυτά που λέτε. Επίση χαιρετίζουμε και την υποχρέωση απόδοση λογαριασμών, ε, κυρίως αυτή που αφορά στην Οδηγία 53, απόδοση λογαριασμών σε τρίμηνη βάση. Αυτό θα οδηγήσει ε, βέβαια ε, στο να υπάρχει μεγαλύτερη επιβάρυνση για τις ε, μικρές επιχειρήσεις, όμως κάτι τέτοιο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ίσως δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να απαγορεύσουμε το asset by asset reporting. Σύμφωνα με το άρθρο 54 θα πρέπει να απαγορεύεται να τίθενται κάποιες ερωτήσεις. Αυτό όμως εξεπερνάει κατά πολύ το στόχο μα και γι' αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Κατά τα άλλα, Για να συνοψίσω, Όσον αφορά την βασική κατεύθυνση που ακολουθεί η συμφωνούμε. Σε ορισμένα θέματα επιθυμούμε να συζητήσουμε περαιτέρω και θα καταθέσουμε και άλλες τροπολογίες. Όμως πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να θέτει ερωτήματα για τα σημαντικά αίτια που οδήγησαν στην κρίση. Και επ' αυτού για τις ασφάλειες θα πρέπει να γίνει μια σε βάθος συζήτηση όπως έγινε και με τις τράπεζες. Πράγματι διαφέρει ο τομέας των ασφαλιών Όμω λοιπόν, όμως και αυτός πλήττεται από την κρίση. Γι' αυτό λοιπόν κατά την άποψή μου έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και ε, χαίρομαι για την συνέχιση της συνεργασίας. Έχουν γιατί πολλά σημεία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για πολύ περιεκτική δουλειά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο που αναφέρθηκε για την τροπολογία 54 από τον κύριο Κίκολτ, ε, που λέει ότι τα κρατημέλη δεν πρέπει να απαιτούν να υποβάλλονται στις υποπτικές αρχές ένας κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων. Ε, αντιλαμβάνουμε την πρόθεση του κύριου Μπάλς, είναι πολύ έντιμη. Αυτό που δεν θέλουμε να έχουμε είναι να έχουμε γραφειοκρατία, και ιδιαίτερα σε, μικρές, σε περίπτωση μικρών εταιριών, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους αυτό που ήδη ψηφίσαμε στην ΙΟΠΑ ε, για την ε, το άρθρο 35, σε ό,τι αφορά τη συλλογή στοιχείων, είπαμε ότι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για να δώσουν τη δυνατότητα στις αρχές να κάνουν τα καθηκόντά τους θα πρέπει να παρέχονται. Και προβλέπουμε ότι η απέτηση πληροφοριών είναι απαραίτητη ε, Γι' αυτό δεν θα ήθελα να υποσκάψω ε, τις εξουσίες των αρχών δηλαδή να μπορούν να ζητούν τι απαραίτητε πληροφορίε από τι αρμόδιες αρχέ. Και οι αρμόδιε αρχέ είναι τα κράτη-μέλη και περιορίζουμε τα κράτη-μέλη σε αυτό τον τομέα τη παροχή πληροφοριών. Δεν νομίζω να είναι η πρόθεση του εισηγητή, αλλά ε, θα μπορούσε έτσι όπω έχει συνταχθεί ε, ιδιαίτερα αν έχουμε να κάνουμε με πάτες, να, να μην δώσει τη δυνατότητα σε αυτές τις αρχές να διεκπαιρέσουν ε, τα καθήκοντά που τους έχουμε αναθέσει. Γι' αυτό, αυτό ε, δεν συνάδει με αυτό που ήδη ψηφίσαμε στις ρυθμιστικές εξουσίες που έχουμε δώσει στις αρχές. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να διορθωθεί με μια πολύ εύκολη τροπολογία. Θα μπορούσα να συνεργαστώ με τον εισηγητή έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και οι δύο προθέσεις για να δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Αλλά ε, πιστεύω ότι το έργο που έκανε ο εισηγητής είναι όπως πάντα πολύ αποτελεσματικό, λεπτομερές και υποστηρίζω ε, τη δουλειά που έχει γίνει για τις οπολογίες μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ, Ζαν Πολ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λίγες παρατηρήσεις θα κάνω αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα συγχαρώ τον Μπούρκαρτ για την εξαιρετική δουλειά που έκανε για ένα τόσο πολύπλοκο θέμα. Προτείνει λύσεις ευφυείς και εύστοχες. Θα ήθελα μόνο δύο θέματα συγκεκριμένα να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, χαιρετίζω τη βούληση που υπάρχει ώστε να έχει πραγματικές αρμοδιότητες η ΟΠΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιθυμεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους σχετικά αφορούμενους τομείς και πιστεύω ότι οι προτάσεις του Μπούκαρτ είναι εξαιρετικέ. Τώρα, αυτό το θέμα της ε, ε, πριμ, αυτής πριμοδότης αντικυκλικής, της ε, μη είναι ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί. Νομίζω ότι θα συζητήσουμε περαιτέρω ε, το θέμα της θέσης σε εφαρμογή θέσης της ε, οδηγίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και το χρονοδιάγραμμα επίσης είναι εξίσου σημαντικό για να είναι σε όλους τους μηχανισμός. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει απαραίτητο να κάνουμε τρία πράγματα για το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα, οι λύσει που θα υιοθετήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι από τεχνική πλευρά οι κατάλληλε, διότι μια καλή νομοθεσία δεν σημαίνει μόνο καλή οργάνωση διοικητική, αλλά πάρα πολύ καλές τεχνικές διατάξεις. Δεύτερον, θα πρέπει αυτό να γίνει έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα, διότι αν έχουμε διάφορε εξαιρέσει και εθνικέ διατάξει, δεν θα κάνουμε τίποτε το σωστό. Ξέρουμε ότι οι σχέσεις με τις τρίτες χώρες είναι σημαντικές, αλλά οι ε, ευρωπαϊκοί κανονισμοί θα πρέπει να είναι για μας πάρα πολύ σημαντικοί σε σχέση με το τι έχουμε να κάνουμε με τρίτες χώρες. Και τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει στην διατύπωση της οδηγίας η καλύτερη δια... δυνατή ποιότητα και να έχουμε κείμενα ευανάγνωστα και που δεν επιδέχονται διτέ ερμηνείε εκ των υστέρων, διότι δημιουργείται ασάφεια και δυσκολία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί διότι μόνον έτσι, αν παρουσιάσουμε ένα πολύ καλό κείμενο με καλά επιχειρήματα, θα ε, πείσουμε και το Συμβούλιο μας ακολουθήσει. Και θα ήθελα να πω το εξής στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να είμαστε σαφεί. Δεν μπορούμε να ζητούμε συγχρόνω να είναι αποτελεσματικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποδοτικό και να βάζουμε ήδη στον εαυτό μα περιορισμού και τροχοπέδι. Ο... Ένα από του νομοθέτε είμαστε κι εμείς. Δεν θα πρέπει να μειώσουμε λοιπόν τις νομοθετικές εξουσίες του Κοινοβουλίου σήμερα κάνοντας αναφορά στο κείμενο Νερόνι, το οποίο αναφερόταν σε μια εποχή που άλλαξε διαπαντός και σε μια κατάσταση τελείως διαφορετική. Επίσης, τα διάφορα κείμενα στα οποία κινδυνεύουμε να πνιγούμε δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς και να έχουμε, επαναλαμβάνω, ε, βανάγνωστα και σαφή κείμενα στα οποία να βασιστούμε. Ευχαριστώ. Μόνο τότε έτσι θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η δουλειά μας. Ο Μπούρκαρτ. Κοιτάξτε, έχοντας ε, κατά νου το χρόνο, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναντέλφου για αυτά ε, που μας είπαν. Νομίζω ότι εκφράστηκαν πάρα πολλές απόψεις ε, και για μένα λοιπόν ε, είναι απόλυτα σαφές ότι τις επόμενες ε, εβδομάδες ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε κυρίως ε, για το θέμα της ε, ισοτιμίας των τρίτων χωρών. Επίσης να ασχοληθούμε με τους εφαρμοστικούς κανόνες και τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Όλα αυτά να διευθυνιστούν και να δούμε λιγάκι και το θέμα του πριμ ρευστότητας. Όσον αφορά στις μεταβατικές διατάξεις, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες να βρούμε κάποια λύση και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι εγκρίνονται περισσότερα δικαιώματα για τον φορέα ΑΙΟΠΑ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μου επισημάνατε κυρία Πρόεδρε ε, και χαίρομαι πάρα πολύ για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει γιατί την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε στο Στρασβούργο με τους σκιώδης και εκεί ε, θα μπορούμε να έχουμε διμερείς ε, επαφές και συζητήσεις όπου όλα αυτά τα θέματα θα συζητηθούν ε, λεπτομερώς. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και νομίζω ότι είμαστε αναμφίβολα σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι 12.30. Και όπως είπα προηγουμένως, το θέμα το 9, η Ευρωπαϊκή Διάσταση των Αθλητισμών, θα συζητηθεί μετά το τέλος της ψηφοφορίας σήμερα το απόγευμα. Θα είστε ούτως ή άλλως εδώ για να ψηφίσετε και σας ευχαριστώ που θα παραμείνετε και μετά. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για όλους που ήταν εδώ και περίμενα να μιλήσουν, αλλά θα επαναλαμβάνω μετά την ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα θα εξεταστεί το θέμα σας αυτό για τον αθλητισμό. Ευχαριστώ λίγο τη συνεδρία.